Πιστεύουμε πως με βάση αυτές τις αξίες ε, περισσότερο έχουμε δύναμη και όχι αδυναμία ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι ο μελλοντικός κανονισμός ε, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ε, είναι, θα αποτελέσει πραγματικά μια μεγαλύτερη ισχύ για την Ευρώπη. Τι πιστεύουμε εμείς για τον κανονισμό αυτό. Από την πρώτη στιγμή εμείς δεν συλλέγουμε δεδομένα. Είμαστε μια μηχανή αναζήτησης που σέβεται την ιδιωτική ζωή. Είμαστε μάλιστα η μόνη μηχανή αναζήτησης πιστεύουμε στην ε, προστασία της ιδιωτικής ζωής εξορισμού και από το σχεδιασμό όπως ζητά το άρθρο 25 του κανονισμού. Το ιστορικό αναζήτησης πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι απόλυτα προσωπικό για απλούς και σαφείς λόγους γιατί το ιστορικό αναζήτησης είναι πολύ ευαίσθητο γιατί λέει, ε, δίνει πληροφορίες για το ποιος είστε, δίνει τις πολιτικές σας ε, πεπιθήσεις, ε, τις σεξουαλικές σας προτιμήσεις, πληροφορίες για τα, έσοδα, για τα εισοδήματά σας, για το, την υγεία σας γιατί ό,τι χρειάζεται να ξέρει κάποιος άνθρωπος σήμερα, κάποιο πρόσωπο, ε, το βρίσκει σε μια μηχανή αναζήτησης. Εμείς λοιπόν προσφέρουμε τις πληροφορίες χωρίς να συλλέχουμε προσωπικά δεδομένα. Η ιδέα είναι πως η ιδιωτική ζωή θα πρέπει να μετατραπεί και από τεχνολογικής άποψη, ώστε να υπάρχουν καλά αποτελέσματα, πάντοτε προτάσσοντας το γεγονός ότι δεν συλλέγουμε ε, στοιχεία ε, προσωπικά. Ε, επί τη βάση λοιπόν του σεβασμού της ιδιωτικής, της προσωπικής ζωής και με, λόγω του ότι συλλέγουμε στοιχεία στο ίντερνετ μπορούμε να κάνουμε τεχνητή νοημοσύνη χωρίς όμως να θέσουμε σε κίνδυνο τα προσωπικά στοιχεία. η τεχνητή νοημοσύνη ε, ότι απαιτεί τα προσωπικά στοιχεία, αυτό είναι μια κατάχρηση. Για να κάνει κανείς τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται πάρα πολλά στοιχεία. Ωστόσο μπορούμε να κρύψουμε το προσωπικό κομμάτι των στοιχείων. Ένα παράδειγμα, αν έπαιρνα τα στοιχεία σας για να κάνω τεχνητή νοημοσύνη για ένα ε, ιατρικό προϊόν, φυσικά θα χρειάζομαι όλα τα στοιχεία για την υγεία σας, αλλά ε, δεν χρειάζεται να ξέρω αν είστε εσείς που υποφέρετε από γρήπη ή ε, ε, θα δώσουμε τη λύση στον ε, γιατρό σας, στον προσωπικό σας γιατρό, αλλά ε, εκείνος μόνο θα γνωρίζει ότι πρόκειται για σας τον ίδιο και για τα δικά σας δεδομένα. Οι προτάσεις για τους χρήστες για το γεγονός ότι τα στοιχεία τους δεν συλλέγονται ή συλλέγονται, εάν ακολουθήσουμε αυτόν τον κανονισμό, συγκεκριμένα πρέπει να εντοπίζονται ε, σε περίπτωση συλλογής και επεξεργασίας. Εμείς θεωρούμε πως αυτό αποτελεί ισχύ για την Ευρώπη και για το ευρωπαϊκό οικοσύστημα. Είναι οι αξίες μας, είναι ευρωπαϊκές αξίες να προστατεύονται οι ε, επιχειρηματίε, γιατί δεν είναι η Ευρώπη κατά των επιχειρήσεων ε, εννοείται, αλλά να προστατεύεται και ο καταναλωτής πρώτα απ' όλα. Η Quant τα πάει πολύ καλά ε, φτιάχνει τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά σεβόμενοι τις υποχρεώσεις για την μη διατήρηση των προσωπικών δεδομένων και σεβόμενοι απόλυτα τον κανονισμό. Για τον απλό λόγο ότι σε σχέση με την επιχείρησή σας και με το μοντέλο της επιχείρησής σας, το επιχειρηματικό σας μοντέλο, η συλλογή δεδομένων, κυρίως ε, τη αγνία των χρηστών, είναι ένας τρόπος μόνο για να πλουτίσει κανείς περισσότερο. Ε, δεν είναι τρόπος αυτός για να κερδίσει χρήματα στο ίντερνετ. Και για να σας δώσω μια μικρή απόδειξη, να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα η Google είπε ότι ο κανονισμός δεν θα την επηρεάσει τόσο για τον απλό λόγο ότι το 80% του κύκλου εργασιών προέρχεται από την προσθήκη λέξεων. Δηλαδή όταν αναζητείτε κάτι, κάνετε να γράφετε μία λέξη, κάνετε ένα κλικ ε, σε αυτή τη λέξη και ε, μετά σας δίνει τα αποτελέσματα. Εμείς δεν χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε αν είστε άνδρας ή γυναίκα, ποια είναι η θρησκεία σας, τίποτα. Και όταν το λέει ο ίδιος, το ίδιο το αφεντικό της Google, να σας πω και εγώ ως αφεντικό της Quant ότι έχει δίκιο. Εδώ και έξι χρόνια το λέω ότι δεν χρειαζόμαστε τα στοιχεία σας για να κερδίσουμε χρήματα. Και σας το λέω σήμερα γιατί τώρα σας λένε ότι χρειάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για να φτιάξουν τεχνητή νοημοσύνη και ότι αυτό θα θέσει πρόβλημα σε σχέση με την τεχνολογία στην Ευρώπη. Εγώ σας το λέω δεν χρειαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για να κάνουμε τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και αν χρειαζόμαστε πάρα πολλά στοιχεία. Ο κανονισμός λοιπόν μπορεί να επιτρέψει στην Ευρώπη να προτάξει τις αξίες της και οι υπόλοιποι ας συμμορφωθούν και ας μην κάνουν τον κόσμο να πιστεύει ότι όσο πιο πολλά στοιχεία συγκεντρώνουν ε, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι. Δηλαδή δεν, μπορείτε δεν χρειάζονται αυτά τα στοιχεία για να εγκαταστήσετε μια, μια εφαρμογή για, το, για τον καιρό. Αυτά το κάνουν για να συλλέγουν ε, τα δεδομένα για περισσότερο κέρδος. Και χρησιμοποιούν το γεγονός ότι δεν ξέρατε ότι θα συλλέξουν αυτά τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτά λοιπόν και έχω να μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις και θέλω όλος ιδιαίτερος να ευχαριστήσω το γαλλικό, την Γαλλική Συνέλευση που χθε το βράδυ υπερψήφισε το άρθρο 17α που αφορά την εφαρμογή την μεταγραφή του κανονισμού αυτού στη γαλλική νομοθεσία σημαίνει ότι όταν ανάβετε το δικό σας κινητό τηλέφωνο, εξορισμού ορισμένοι γίγαντες πληρώνουν για να είναι εγκατεστημένοι εξορισμού. Και τώρα όμως ε, θα έχετε εσείς την επιλογή γιατί έχει αφαιρεθεί η λέξη economy από την, από το άρθρο. Οι χρήστες λοιπόν από σήμερα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ε, τη μηχανή αναζήτησης που θα εγκαταστήσουν στο κινητό του τηλέφωνο. Μπορεί να είναι ο φίλος μας ο Αμερικάνος, μπορεί όμως να είμαστε εμείς. έχετε την επιλογή. Ο, ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ ε, κύριε. Θα προχωρήσουμε τώρα στην κυρία Μαρνό. Με μικρόφωνο παρακαλούμε να ανοίξει το μικρόφωνο. Ευχαριστώ αγαπητέ κύριε Πρόεδρε αξιότιμες κυρίες και κύριοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να ομιλήσω στη σημερινή σας εκδήλωση για, την, ε, για τις επιπτώσεις της εφαρμογής του GDPR στην ε, ε, μελλοντική εξέλιξη ψηφιακής οικονομίας. Προέρχομαι από το Γερμανικό Ινστιτούτο Ερευνών και ιδίω ασχολούμαι με το σημείο όπου τέμνεται η τεχνολογία με την νομοθεσία και το λέμε και privacy by design, καθώς και λύσεις για την ψηφιακή τεχνολογία. Κυρίως θα αναφερθώ στην πρόοδο της έρευνας σχετικά με τον GDPR, δηλαδή τον βασικό κανονισμό, και με τις επιπτώσεις του. Ο κανονισμός βασίζεται στην τεχνολογική εξέλιξη. Παραδείγματα, η οδηγία βασιζόταν κυρίως στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Όμως ο κανονισμός έχει μια βάση στην ανάλυση του κινδύνου και τον ενδιαφέρει κυρίως το πώς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία απαιτούν μέτρα και ιδίω το άρθρο 25 και το άρθρο 32 που ζητούν από τον ελεγκτή των δεδομένων να εξετάζει σε ποια τεχνολογία βασίζονται και ποια τεχνικά μέτρα είναι αναγκαία να εφαρμοστούν. Εκτός αυτού, ο κανονισμός ορίζει ότι με την εφαρμογή ορισμένων τεχνολογικών μέτρων η επεξεργασία δεδομένων μπορεί να τεθεί και εκτός πεδίου εφαρμογής εν μέρη ή και εξ ολοκλήρου. Και η αιτιολογική σκέψη 26 λέει ότι ο GDPR δεν εφαρμόζεται σε ανώνυμα δεδομένα. Το άρθρο 11 επιτρέπει στον επόπτη ή μάλλον στον ελεγκτή να, ελέγχει, να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα εφόσον δεν επιτρέπουν αυτά να ε, διαπιστωθεί ποιο είναι το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτό λοιπόν οριοθετεί, αυτά μάλλον οριοθετούν και το πεδίο της έρευνας που διεξάγω σχετικά με το που βρίσκεται η τεχνολογία, αυτή τη στιγμή και η τεχνολογία ασφάλειας μεταξύ αυτών. Οι τεχνολογίες ενίσχυσης του προσωπικού χαρακτήρα των δεδομένων από τότε που εγκρίθηκε ο κανονισμός το 2016, εγώ έχω προσωπικά δει μια τεράστια αύξηση ενδιαφέροντος για αυτού του είδους τις τεχνολογίες, privacy enhancing, καθώς και την επιστημονική πρόοδο των τεχνολογιών αυτών, την μεγάλη αύξηση δημοσιευμάτων, εκδηλώσεων, σχετικών διαλέξεων κλπ. Παραδείγματα. Πρώτα, εκεί που ενδιαφέρομαι εγώ εδώ για την αναλογικοποίηση δηλαδή και που είναι ε, και μέσα σε ένα πλαίσιο ε, όλο και περισσότερων εξελίξεων εμείς βλέπουμε κάπου όπου η αναλογικοποίηση δεν είναι επαρκή και τα υποκείμενα των ε, δεδομένων είναι δυνατόν να εντοπιστούν. Όμως η επιστήμη έχει ε, κάνει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια και υπάρχουν νέες τεχνικές ανωνυμοποίησης όπως η preferential και ε, από το 2016 συνάδελφοί μου και εγώ αντιμετωπίζουμε αύξηση ενδιαφέροντος όχι μόνο για τις επιστημονικές δημοσίευσεις αλλά και από πλευράς επιχειρήσεων που θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας για να χρησιμοποιήσουν τις πιο προηγμένες τεχνολογίες εχμής για την ανωνυμοποίηση και να εφαρμόσουν τις τεχνικές αυτές στα πραγματικά τους προϊόντα που θέτουν δηλαδή σε, στην αγορά. Αυτό το βλέπουμε, την τη ζήτηση μόνο αυτή τη βλέπουμε μόνο από πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υστερούν κατά πολύ. Θα ήθελα λοιπόν να δω το ενδιαφέρον αυτό για τεχνολογίες εχμής να φτάσει να απασχολήσει μέχρι και τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και να έχουν μεγαλύτερη ε, ε, ανάγκη και ζήτηση να συνεργαστούν με του ερευνητέ και επιστήμονε. Άλλο παράδειγμα είναι ότι οι απαιτήσει του κανονισμού συζητούνται παντού και επηρεάζουν και τα θέματα των μεγάλων ε, διοργανώσεων που ασχολούνται με την ασφάλεια επιστημονικών συνεδρίων κλπ. Όλοι γνωρίζετε περί της τεχνολογίας blockchain για την οποία όλοι συζητούν πλέον και συζητείται πάρα πολύ ως μια ενδεχόμενη λύση για οποιαδήποτε σχεδόν πτυχή της εξέλιξης από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορείτε να σκεφτείτε. Όμως οι διαδικασίες κρυπτογράφησης έρχονται σε αντίθεση με την προστασία δεδομένων. Θα πρέπει να είναι μια πτυχή του ίδιου του συστήματος, δηλαδή να υπάρχει το δικαίωμα λύθης για το πρόσωπο, να μπορεί να ζητήσει να διαγραφούν τα δεδομένα του και να λησμονηθεί από αυτόν που ελέγχει τα δεδομένα. Συνάδελφοί μου έχουν προτείνει τα τελευταία χρόνια ορισμένε ενδεχόμενες λύσεις ώστε στην blockchain να μπουν νέες κρυπτογραφικές δυνατότητες η κοινότητα των όσων ασχολούνται με την ασφάλεια γνωρίζει καλά τι συμβαίνει με τον κανονισμό GDPR. Παρόλο που αντιμετωπίζουν κάποιε προκλήσει ό,τι αφορά την ερμηνεία του νομοθετικού κειμένου και να τι μεταφράσουν δηλαδή σε πράγματα τα οποία να είναι δυνατόν να υλοποιηθούν από την τεχνολογία, προσπαθούν ακριβώ λοιπόν αυτό να κάνουν. Θα δείτε στι σημειώσει που έχω δώσει και του σχετικού συνδέσμου για τα έγγραφα αυτά που είναι δημοσιευμένα στο διαδίκτυο. Εγώ είμαι πολύ θετική απέναντι στις επιπτώσεις του GDPR. Ωστόσο βλέπω να υπάρχουν ακόμα κάποιες προκλήσεις. Προκλήσεις που αναφέρονται σε κάθε ομάδα ενδιαφερομένων και τους ερευνητές και τις εποπτικές αρχές και τις αρχές προστασίας δεδομένων ακόμα και τους νομοθέτες. Θέλω λοιπόν να τονίσω ορισμένες από τις προκλήσεις αυτές και πολύ ευχαρίστως να τις συζητήσουμε αν θέλετε μετά χρειαζόμαστε περισσότερη διακλαδική έρευνα και χρειαζόμαστε και τυποποιημένες διαδικασίες για την αξιολόγηση του κινδύνου. Γιατί χρειαζόμαστε μια εργαλειοθήκη για την ε, ανάλυση των τεχνολογιών. Δεν χρησιμοποιούμε ούτε καν την ίδια ορολογία. Χρειάζεται να γίνουν διακλαδικές λοιπόν προσπάθειες για να μεταφράσουμε τις νομοθετικές απαιτήσει σε τεχνολογία. Τις privacy requirements σε τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα sprint coding. Έχουμε ανάγκη και από διακλαδική συνεργασία για την, αντιμετώπιση και τον, για την ανάλυση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το άτομο. Χρειαζόμαστε μια εναρμονισμένη λοιπόν ερμηνεία των TPA σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα ήθελα να δω και κάποιες βέλτιστες πρακτικές και κατευθυντήρες γραμμές από τους DPA σε πολλά άρθρα του ο κανονισμό ζητεί να ληφθεί υπόψη το state of the art, δηλαδή το που ακριβώ βρίσκεται η τεχνολογία. Αλλά δεν είναι σαφέ ποιο είναι αυτό, ακόμα και του ερευνητέ δεν είναι σαφέ. Δεν υπάρχουν και συγκεκριμένοι ορισμοί, ευσύνοπτοι συγκεκριμένοι ορισμοί. Και αυτό εν τέλει θα οδηγήσει να κρίνεται αυτό το state of the art αναπερίπτωση από τα δικαστήρια που θα καλούνται να ε, εγκύψουν στις υποθέσεις DPA. Εγώ θα ήθελα να είναι εκ των προτέρων γνωστές οι κατευθυντήρες αυτές τις γραμμές. Ορισμένες DPA το κάνουν αυτό από την αρχή και χρειάζεται εναρμόνισή τους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηριχτούν αυτοί που ελέγχουν τα δεδομένα και αυτοί που τα επεξεργάζονται θα πρέπει να έχουν έναν αριθμό βέλτιστων πρακτικών πάνω στι οποίε να μπορούν να προσανατολίζονται. Και θα είναι σωστό επίση να υπάρχουν διεθνή πρότυπα για το privacy engineering για να γνωρίζουμε πού βρίσκονται το state of the art σε θέματα ασφάλεια. Και αυτά να τα αποφασίζουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, από του ε, χρήστε μέχρι του επόπτε. Πώ μπορούν ε, να υλοποιηθούν αυτές οι βέλτιστες πρακτικές. Αυτά για παράδειγμα και στον ε, τομέα της υγείας. Άρχισαν να κάνουν μια προσπάθεια ζητώντας παραδείγματα των πρακτικών σε εφαρμογές για θέματα υγείας. Εγώ αναμένω να δω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εργασιών αυτών, γιατί η ηλεκτρονική υγεία χρειάζεται απαραίτητα τις βέλτιστες πρακτικές και privacy by design. Υπάρχουν τώρα και οι προκλήσεις για τους νομοθέτες, τουλάχιστον από την άποψη του ερευνητού ή της ερευνήτριας. Σε ό,τι αφορά την τεχνολογική εξέλιξη και την προστασία δεδομένων. Διότι έχω δει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες μέλη νομοθετικές πρωτοβουλίες για την έγκριση αυστηρότερης νομοθεσίας κατά της κατάχρησης των δεδομένων και ιδίως ό,τι αφορά το κυβέρνο έγκλημα, ξεκινώντας από την απαγόρευση της ε, μη εγκεκριμένης χρήσης ε, ηλεκτρονικής τεχνολογίας μέχρι και άλλα θέματα προστασίας δεδομένων και μάλιστα και στην διάσκεψη των Γερμανών TPA που ζήτησαν από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να προτείνει ποινικό δίκαιο που να απαγορεύει την ε, διασύνδεση για την χρήση ορισμένων ιατρικών δεδομένων. Εγώ θεωρώ ότι οι νομοθέτες πρέπει να σκεφτούν ποιοι είναι οι κίνδυνοι αυτών των νομοθετικών πρωτοβουλειών. Διότι η έρευνα, οι ερευνητές μάλλον, χρειάζονται και κάποια ελευθερία χρειάζονται την ελευθερία να μπορούν να προσβάλλουν τα συστήματα για να δουν πού είναι τα αδύναμα σημεία τους, πού βρίσκονται τα τροτά σημεία των συστημάτων ηλεκτρονικής εξεργασίας δεδομένων και πού βρίσκονται οι κίνδυνοι για την προσωπική σφαίρα. Αν μου επιτρέπετε να δώσω λίγα ακόμα παραδείγματα. Οι συνάδελφοί μου εντόπισαν ότι αυτό που πίστευαν οι ερευνητέ ότι τα επεγενετικά δεδομένα είναι στην πραγματικότητα ανώνυμα δεν είναι αληθέ. Διότι ναι μεν αλλάζουν διαρκώς, αλλά παρόλα αυτά επιτρέπουν τον εντοπισμό του υποκειμένου των δεδομένων. Έχουμε συνεργαστεί με το Αντικαρκυνικό ε, Ίδρυμα Ερευνών για να δούμε Και αν δεν υπήρχε η δυνατότητα διασύνδεσης που πρόβλημα αρχικά ο νόμος, ποτέ δεν θα είχαμε μπορέσει να εντοπίσουμε αυτό το τρώτο σημείο. Άρα, επιτρέψτε στους ερευνητές να αναλαμβάνουν κάποιους κινδύνους για να μπορούν να εντοπίζουν τα τρώτα συστήματα, των, τα, τα, σημεία μάλλον των ηλεκτρονικών συστημάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη θαυμάσια αυτή παρέμβασή σας. Τέλος, ο κ. Μπράιταρτ. Ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ε, κυρίε και κύριοι, πρώτα απ' όλα σα ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να είμαι εδώ σήμερα. Όπω είπα πριν, σε 10 μέρε η αναμονή τελειώνει και η πρώτη φάση μεταρρύθμιση του νομικού, μεταρρύθμιση του πλαισίου ολοκληρώνεται. Έχω εμπλακεί στη συζήτηση από το 2011 πρώτα ως ε, διεθνής ε, λειτουργός αρμόδιος για τα θέματα αυτά στην Ολλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων και τα τελευταία χρόνια στην νήμητη μιας, εταιρεία, μιας εταιρείας έρευνας και λογισμικού. Όπως ήδη ακούσατε σήμερα, ο κανονισμός αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικό νομοθέτημα και εδώ και χρόνια όλοι οι αρμόδιοι για αυτά τα ζητήματα μόνο τον κανονισμό αυτό συζητούν και πολλοί οργανισμοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί δουλεύουν σκληρά για να μπορέσουν να συμμορφωθούν μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Βεβαίω, δεν καθόταν όλοι τα τελευταία δύο χρόνια, ούτε ξύπνησαν όλοι τον τελευταίο μήνα. Αλλά πράγματι, τις τελευταίες εβδομάδες βλέπουμε ότι όλο και περισσότερες εταιρείε ε, συνειδητοποιούν ότι υπάρχει ο κανονισμός και κάτι πρέπει να γίνει. Η συμμόρφωση λοιπόν με τον κανονισμό είναι κάτι το οποίο εύκολα λέγεται, αλλά δύσκολα γίνεται. Αυτό βεβαίως μπορεί να προξενεί έκπληξη γιατί κατ' ουσίαν μιλάμε για μια μετεξέλιξη και όχι μια επανάσταση. Αλλά όσοι το έπαιρναν σοβαρά ήδη από την οδηγία του 1995 και την εθνική νομοθεσία και αυτοί θα έχουν ε, σοβαρή προσπάθεια να κάνουν. Θα πρέπει να αναθεωρηθούν συμφωνίες προς τα Προστασία και επεξεργασία δεδομένων, πολιτικέ ε, και διαδικασίε. Ε, μέχρι πρόσφατα αυτά ήταν ε, κυρίω δουλειά που έκανε ένα άτομο ή μια μικρή ομάδα ατόμων που κατά κανόνα δεν έκαναν και όλη την ώρα αυτό. Εδώ πέρα λοιπόν έχει επέλθει μια αλλαγή της νοοτροπίας σε πολλούς οργανισμούς και όσον αφορά την ετελική κουλτούρα κατά την άποψή μου η αλλαγή αυτή οφείλεται στην υποχρέωση λόγοδοσίας που αναφέρεται στα άρθρα 5 και 24 του κανονισμού οι οργανισμοί τώρα θα πρέπει να έχουν ενσωματώσει την προστασία δεδομένων στην επιχειρησιακή τους λειτουργία και να μπορούν να αποδείξουν την συμμόρφωσή τους με τις ουσιαστικές διατάξεις του κανονισμού σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού τους. Δηλαδή το να αποτελεί πλέον η υπόθεση αυτή, η υπόθεση ενός ατόμου που θα βρίσκεται στο τμήμα το νομικό ή της συμμόρφωσης πλέον δεν αρκεί. Πρόκειται επίσης και για μια άλλη μεγάλη αραγή η οποία έχει επέλθει. Υπήρχε εξειδικευμένο λογισμικό επί σειρά ετών για τα διάφορα τμήματα μεγάλων εταιριών από το λογιστήριο μέχρι το τμήμα προσωπικού και τώρα αναπτύσσεται και ανάλογο λογισμικό για αυτόν τον τομέα. Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε αυτόν τον ε, τομέα όσον αφορά της βάσης δεδομένων και αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στα 770 νομοθετήματα για την ιδιωτική ζωή παγκοσμίω. Με τα οποία βέβαια πρέπει να προσαρμόζονται πολλέ εταιρείε. Εδώ πέρα λοιπόν έχουν αναπτυχθεί νέε λύσει λογισμικού, έτσι ώστε οι εταιρείε να μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα, να γίνονται αυτοματοποιημένε αξιολογήσει αντικτύπου και να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν αυτέ ω νομική βάση επεξεργασία δεδομένων. Αν εξετάσετε έναν κανονισμό λοιπόν από τη σκοπιά τη καινοτομία, αναγκάζει εμά και του ανταγωνιστέ μα να βρούμε νέε ιδέε για να μπορέσουν να συμμορφωθούν οι οργανισμοί ευκολότερα. Λέω ευκολότερα, γιατί η συμμόρφωση με την προστασία των δεδομένων δεν είναι ποτέ εύκολη, ούτε είναι κάτι το άσπρο και μαύρο. Ο βασικό μα στόχο δεν είναι να υπάρξει μια πλήρης αυτοματοποίηση και δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Καθώς η νομοθεσία αυτή βασίζεται σε κανόνες και πάντα θα απαιτεί μια ανθρώπινη αξιολόγηση. Αλλά το έξυπνο λογισμικό το οποίο βασίζεται σε πάρα πολλές ώρες έρευνας μπορεί να απλοποιήσει αυτή την διαδικασία. Ο δικός μας ο κλάδος έρευνας παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις νομοθετικές εξελίξεις, ε, την ομολογία και τις σχετικές αποφάσεις και αυτό μας επιτρέπει να φτιάξουμε κάποιες βάσεις δεδομένων πραγμάτων που επιτρέπονται και απαγορεύονται, από τις οποίες μπορούν να ωφεληθούν οι συνδρομητές μας. Αυτό σε συνδυασμό με την σχετική υπηρεσία που θα αναπτυχθεί σε κάθε εταιρεία θα, υπάρχει, θα δώσει τη δυνατότητα στις εταιρείες να προσαρμοστούν χωρίς να υπάρξει ανάγκη εκτεταμένης εκπαίδευσης. Ειδικά το τελευταίο έτος αναπτύξαμε κάποιες νέες μεθοδολογίες για να στηρίξουμε την ε, συμμόρφωση περιλαμβανομένων και εργαλείων για λογοδοσία και ιδιωτικότητα ήδη από τη φάση του σχεδιασμού. Έτσι μπορούν να βρεθούν τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα εκείνα τα οποία θα επιτρέψουν στις εταιρείε να χειριστούν τα προσωπικά δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους. Έτσι θα πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται την προστασία των δεδομένων από νωρί, να την ενσωματώσουν δηλαδή στο σχεδιασμό των διαδικασίων τους. Η διαδικασία αυτή επίσης καθιστά ευκολότερο το να μπορεί κάποιος να πει το πώς διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων από τεχνικά μέτρα όπως κρυπτογράφηση και περιορισμού στην πρόσβαση μέχρι μέτρα εντός του οργανισμού οι βασικοί μας πελάτες είναι οργανισμοί οι οποίοι θέλουν να έχουν μια υπεύθυνη προσέγγιση στην ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων και βεβαίως τους στηρίζουμε σε αυτό το στόχο. Έχουμε λοιπόν μία βάση σύγκρισης ε, την οποία χρησιμοποιούν οι πελάτες μας και γνωρίζουμε πως όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι σημαντικοί και για αυτούς. Να σας πω κάποιους αριθμούς. 48 πελάτες μας έχουν λάβει μέρος σε μία συγκριτική αξιολόγηση για να δουν πώς θα πηγαίνουν με βάση συγκεκριμένες δραστηριότητες διαχείρισης της ιδιωτικότητας. Δηλαδή, για δραστηριότητες ε, οι οποίες έχουν ήδη εφαρμοστεί ή είναι στην φάση της εφαρμογής, ε, είτε είναι στην φάση του σχεδιασμού ή είναι απλά κάτι το επιθυμητό. Αλλά ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Και σε κάποιες ε, επίσης περιπτώσεις δεν ισχύουν ε, αυτές οι διατάξεις παραδείγματος χάρη αν δεν επεξεργάζονται δεδομένα ανηλίκων δεν υπάρχει και ανάλογη δραστηριότητα. Να σας δώσω λοιπόν τα πρώτα αποτελέσματα. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα ενσωμάτωση από τον σχεδιασμό ήδη. 23%, 23 των οργανισμών το κάνουν ήδη αυτό, 48% είναι κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη και 27% των οργανισμών αυτών είναι ακόμα στην φάση όπου είναι Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Και σε 2% των περιπτώσεων δεν ισχύει, δεν υπάρχει τέτοια απέτηση. Όσον αφορά τώρα τις αξιολογήσεις αντικτύπου, βλέπετε πως κανείς δεν λέει ότι αυτό δεν έχει σημασία. 37% των εταιριών ε, το ε, λένε 23% με λένε ότι είναι κάτι το επιθυμητό, 37% το έχουν εφαρμόσει και 40% λένε ότι είναι εν εξελίξη. Αν δούμε παρακάτω, βλέπουμε ότι η τήρηση μητρώου τέτοιων δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων επίσης βρίσκεται σε καλό δρόμο. 21% λένε πως το έχουν ολοκληρώσει, 62% είναι αυτή τη στιγμή στην διαδικασία υλοποίησης και 17% λένε θέλουμε αλλά δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Και εδώ πέρα θεωρώ πως οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες θα παραμείνουν σε μια διαδικασία υλοποίηση, γιατί δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ αυτή η διαδικασία, θα ενημερώνεται συνεχώ. Με βάση και την κατεύθυνση που θα δίνει η ομάδα εργασία του άρθρου 29 τέλο, τα τελευταία στοιχεία που θέλω να σα ε, δώσω, όσον αφορά την κρυπτογράφηση προσωπικών δεδομένων. Ήδη 62% των ε, οργανισμών ε, που είναι πελάτες μας το έχουν εφαρμόσει και 17% είναι στην διαδικασία υλοποίησης. Θα ήθελα λοιπόν να πω πως η συμμόρφωση με τον οργανισμό δεν απαιτεί πάντα λογισμικό αντιθέτως. Για μικρούς οργανισμούς ή για όσους έχουν απλές τέτοιες λειτουργίες σε λίγες χώρες, συχνά αρκεί ένα λογιστικό φύλλο. Αυτή τη στιγμή όμως οι διαδικασίες αυτές αποκτήσουν μεγάλο όγκο ή περιπλοκότητα λόγω της φύσης των δεδομένων ή των αριθμό των χωρών όπου δραστηριοποιείται κάποιος, το λογισμικό αυτό θα αποδείξει την αξία του. Όπως δήλωσε πρόσφατα και ένας ε, αρμόδιος ε, επόπτης προστασίας προσωπικών δεδομένων, 25 Μαΐου είναι απλά το τέλος της αρχής του κανονισμού. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια και αναμένουμε την συνεργασία με τους πελάτες μας, ε, τις ρυθμιστικές αρχές και τους νομοθέτες για να διασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και αναμένω τις ερωτήσεις σας. Um, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, συνάδελφοι, θα ακούσουμε τις δικές σας ερωτήσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο κ. Σταγιάννη, έρχεται. Θέλει και εκείνος να απευθύνει ένα χαιρετισμό, να πει δύο λόγια. Και όταν έρθει, αν δεν σας πειράζει, θα ήθελα να του δώσουμε τον λόγο. Δεν έχει έρθει όμως ακόμα. Οπότε μπορούμε να ακούσουμε τις πρώτες ερωτήσεις. Ο κύριος Σπολίτης από την Λετωνία ε, έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για τις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Έχω ερωτήσεις προς την κυρία Μαρνάου αλλά και προς τον κύριο Λεάνδρη. Κύριε Λεάνδρη, σας ευχαριστώ που μας είπατε τι έκανε η Γαλλία νομοθετώντας και μεταγράφοντας το νέο κανονισμό. Μιλώντας για τις προκλήσεις, αυτό δεν αφορά μόνο τους αλγορίθμους, αυτό έχουμε σήμερα, αφορά αυτό και το μέλλον. Σε προηγούμενες ε, εισηγήσεις ακούσαμε πως υπάρχουν πολλά πράγματα που είμαστε πίσω λόγω του ότι η τεχνολογία προχωρά τόσο γρήγορα και η έρευνα είναι τόσο ε, γρήγορη επίσης. Αν μιλάμε λοιπόν για τεχνητή νοημοσύνη, εσείς θα έχετε να προτείνετε κάτι ε, που πρέπει να κάνουμε εμείς οι νομοθέτες, ας πούμε χρειαζόμαστε περισσότερους μηχανικούς καλύτερη βασική παιδεία στα σχολεία. Τι άλλο, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ε, κατάσταση. Κυρία Μαρνα, μιλήσατε για προκλήσεις ιδιαίτερα για την ιατρική έρευνα και τις ε, συνδέσεις με τα δεδομένα και μας δώσατε παραδείγματα από τη Γερμανία. Και αυτό με έκανε να σκεφτώ ότι έχουμε φτάσει ένα, το δίλημα του νυχτοφύλακα στον ε, κλασικό φιλελευθερισμό. Μα ζητάτε να εμπιστευτούμε τους ε, ερευνητέ, ενώ ταυτόχρονα ως νομοθέτες οι, κα, οι καταναλωτές, οι, πολίτες ζητούν προστασία των δεδομένων του. Πώ το λύνουμε αυτό. Είδαμε τι έγινε με το Brexit, είδαμε τι έγινε με τις Αμερικανικέ εκλογές το 2016. Εμείς εντωμεταξύ πώ μπορούμε χωρίς να τα κάνουμε όλα θάλασσα, να, δώσουμε, να, να, να, σας δώσουμε την ευθύνη να τα διορθώσετε αυτά, ενώ ταυτόχρονα θα ε, ε, δώ προσφέρουμε και την προστασία των μεγάλων μεταδεδομένων. Σας ευχαριστώ. Θα ακούσουμε ε, διάφορες ερωτήσεις. Ο κύριος Τσέκ από την Σλοβενία την θέση 147. Μάλιστα. Εγώ συμφωνώ με τον συνάδελφο που μόλις πήρε το λόγο. Όμως ακριβώς γι' αυτό χρειαζόμαστε την πολιτική, έναν ε, λογικό και ε, κριτικό μάτι ε, που να μπορέσει να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Εμένα βρίσκει σύμφωνο η θέση της Γαλλίας. Η Quant είναι μία, ένα παράδειγμα σύμμορφο προς το άρθρο 25 στην πρώτη συνεδρία, νομίζω, η Πολωνή συνάδελφό σα είπε ότι δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε του ανθρώπου να χρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Μπορούμε μόνο να αναπτύξουμε εναλλακτικέ. Και αυτή εδώ είναι μια εναλλακτική. Στη Γαλλία γίνεται λόγο και για το ίντερνετ των πραγμάτων. Για παράδειγμα, Έχουμε την ε, περίπτωση των αποβλήτων. Να έχουμε μια εφαρμογή για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς λειτουργεί το σύστημα. Θα πρέπει δηλαδή εμείς οι πολιτικοί να γνωρίζουμε ποια είναι τα απαραίτητα δεδομένα. Ε, εφόσον μας τα ζητήσει η ε, βιομηχανία. Χρειαζόμαστε όλα αυτά για να μπορέσουμε, μπορέσει να λειτουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη και πρέπει να ανταποκριθούμε. Έπειτα, ε, ο Γάλλος ε, συνάδελφος είπε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τις μικρομεσαίες. Έχουμε όμως συνεταιρισμούς, γεωργικούς συνεταιρισμούς. Πρέπει να προωθήσουμε και αυτούς τους συνεταιρισμούς όπου συγκεντρώνονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού αυτές τις προκλήσεις. Μια ερώτηση προς τον κύριο της Quant. Επί τη βάση της δικής σας εμπειρίας, πώς βλέπετε εσείς το ίντερνετ των πραγμάτων στην κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης ή της ανωνυμοποίησης των, δεδομένων. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, μου επιτρέπετε να κάνουμε μια παύση γιατί με μεγάλη μου χαρά πρέπει να σας πω ότι μόλις ήρθε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Αντώνιο Ταγιάννη, που εξέφρασε μέγα ενδιαφέρον στις εργασίες ε, της Επιτροπής μας ιδιαίτερα για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων, για αυτό το τόσο σημαντικό τομέα και ζήτησε να ε, μπορέσει να πάρει το λόγο για ε, λίγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που ήρθατε και παρακαλώ έχετε αμέσως το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Αγαπητοί συνάδελφοι από το Ευρωκοινοβούλιο και από τα Εθνικά Κοινοβούλια, συνάδελφοι, είμαι ευτυχής που είμαι σήμερα εδώ για να παρακολουθήσω αυτήν την διακοινοβουλευτική διάσκεψη για την προστασία των δεδομένων. Οι δέσμοι των μέτρων για την προστασία των δεδομένων αποτελεί μεγάλο ορόσημο, καθώς θα θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Είναι ένα πρώτο τέτοιο παράδειγμα παγκοσμίω. Είμαι πεπισμένος ότι μετά από τόσα χρόνια διαπραγματεύσεων, οι αρμόδιοι διαπραγματευτές βρήκαν την ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών. Ο κανονισμός αυτός αρχίσει να ισχύει σε 10 μέρες ακριβώς. Στις 25 Μαΐου ένα σύνολο ε, ενιαίο κανόνων θα αρχίσει να ισχύει για όλους τους πολίτες και θα εναρμονίσει την προστασία των πολιτών στην Ένωση και θα παρέχει νομική βεβαιότητα για τις επιχειρήσεις. Η πρόσφατη υπόθεση του Facebook μας δείχνει πόσο επίγον είναι να ανακτήσουμε τον έλεγχο επί των ψηφιακών πλατφορμών για να προστατεύσουμε την ιδιωτική μας ζωή οι γίγαντε του δικτύου θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τα δεδομένα μα, αλλά και για το τι δημοσιεύουν συμπεριλαμβανομένων των ψευδών ειδήσεων και του παρανόμου περιεχομένου. Η ελευθερία ε, πάει χέρι-χέρι με την ευθύνη, την ε, υπευθυνότητα. Είμαι ευτυχή που η Επιτροπή σας ζήτησε την να διοργανώσει από την αρχή του Ιουνίου ένα σύνολο ακροάσεων με τους ε, ενδιαφερόμενους φορείς. Αυτές οι ακροάσεις θα προσφέρουν στα μέλη της ΛΥΜΠΕ, της ΑΦΚΟ, της Τζούρι και της Ήτρε την ευκαιρία να ε, κάνουν ε, μία ανάλυση του σκανδάλου του Facebook και με εστιασμό στο, στον δυνητικό αντίκτυπο της διαδικασίας έδωσης στην Ευρώπη. Έχουμε καλέσει και τον κύριο Τζούκερμπεργκ στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε καλέσει όλους τους ειδικού του Facebook. Δουλεύουμε σκληρά για να επιτύχουμε μια συμφωνία με τον κύριο ε, Ζούκερμπεργκ ώστε αυτό να έρθει ενώπιον του Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου διότι θέλουμε να μάθουμε την ιστορία του Facebook για τη διάρκεια του, ε, κατά τη διάρκεια του Brexit, κατά τη διάρκεια των εκλογών και θέλουμε να δρομολογήσουμε μια καλή προεκλογική εκστρατεία πριν τις επόμενες ευρωεκλογές που προβλέπονται για το 2019 η συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι κρίσιμη, ε, πολύ σημαντική εφόσον θέλουμε να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό νομίζω πως η συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και η ΜΟΝ με είναι πολύ σημαντική για το μέλλον εγώ υποστηρίζω εντόνω τη συνεργασία μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Γι' αυτό και η σημερινή μέρα είναι ε, πολύ σπουδαία για την περάσπιση της ελευθερίας μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε στις Βρυξέλλες και στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο Πρόεδρος Μωράε, σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σα σε αυτή την Επιτροπή και για την υποστήριξή σα σε αυτή την νομοθεσία. Ο κύριος Μωράης είναι εξαιρετικός πρόεδρος. Ε, είναι εδώ και ο εισηγητής, ο κύριος Άλμπρεχτ, οπότε είναι ιδανική η κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καλή, καλό σας απόγευμα. So, colleagues, that's the kind of interruption we quite like in this committee. διακοπές μας αρέσουν βεβαίως. Στην Επιτροπή μας είχαμε δύο εξαιρετικές ερωτήσεις ε, από συναδέλφους. Ε, θα συνεχίσουμε λοιπόν. Έχουμε τώρα τον κύριο ε, Ράιο από την Ισπανία. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η κυρία Μαρνάου έθεσε σε ένα ζήτημα που εγώ θεωρώ κέριο. Είναι ο αντίκτυπος του κανονισμού στο πλαίσιο της έρευνας και κυρίως της βιοιατρικής έρευνας. Στην Ισπανία αυτό ήταν ένα θέμα το οποίο προκάλεσε πολλές συζητήσει και αντιδράσεις από πλευράς του ιατρικού τομέα έναντι των πρώτων νομοθετικών πρωτοβουλειών της κυβέρνησης στην προσπάθεια να προσφέρει ε, ρυθμίσεις. Το θέμα είναι κατά πόσο δηλαδή αυτός ο κανονισμός ε, ορθώνει εμπόδια στην ε, ανάπτυξη της έρευνας. Από ό,τι φαίνεται όχι. Όμως ε, το ο κανονισμός επιτρέπει στην εθνική νομοθεσία, επιτρέπει εξαιρέσεις από πολλές εγγύσεις και μπορεί βεβαίως να συμβεί οι χώρες μέλη να, αναπτύξουν, να αναπτυχθούν να αναπτύξουν μάλλον ε, νομοθετικές διατάξεις ε, που θα είναι περιοριστικές ε, για τον ερευνητικό τομέα και κυρίως για την βιοιατρική. Θα θέλαμε λοιπόν να γνωρίζουμε ποια είναι η εντύπωση των εισηγητών μας και ποιες είναι οι εμπειρίες από τις υπόλοιπες χώρες. Γιατί στην Γερμανία ε, περιλαμβάνει σχετική νομοθεσία ε, συγκεκριμένες διατάξεις για την βιοιατρική έρευνα, ε, αλλά δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Πολύ θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε τι συμβαίνει με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Κουπρίβα, Τσεχική Δημοκρατία. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Στην ε, πατρίδα μου, την ψυχική Δημοκρατία, είχαμε και εμείς αυτά τα αρχικά προβλήματα. Έπιασε τον κόσμο μια σχετική ιστερία ότι δεν υπήρχε καμιά μεθοδολογία, ότι η εθνική νομοθεσία δεν ήταν έτοιμη, δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής, η αρχή ε, προστασίας δεδομένων δεν είχε ξεκάθαρες κατευθυντήρες γραμμές και ξαφνικά πάρα πολλοί εμφανίστηκαν που ήθελαν να, δίνουν, να παρέχουν συμβουλές. Εμείς πάντω είπαμε στις μικρές και σε επιχειρήσεις, μη φοβάστε, εάν τηρήσετε τα όσα προβλέπει η νομοθεσία έως τώρα, δηλαδή δεν εκδίδεται ε, ε, έγγραφα με ε, συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα, δεν θα έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Πρόκειται για ένα είδος ε, καινοτομία βέβαια και για τους πολίτες. Και ε, άρχισε η συζήτηση και συνεχίζεται και διεξάγεται και αρχίζουν να συνειδητοποιούν οι πολίτες ορισμένα προσωπικά δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικά και ότι θα πρέπει να προσέχουν τι τα κάνουν. Για παράδειγμα, επίσης, να προσέχουν ας πούμε, τι αναγράφεται στις, στα ατομικά δελτία ταυτότητάς τους. Τονίζουμε δηλαδή ότι ε, δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να προσέχουν και οι ίδιοι πολίτες. Δεν μπορούν να διαθέτουν τα προσωπικά τους δεδομένα ε, χωρίς ε, να προσέχουν τι ακριβώς κάνουν. Και βεβαίως να γνωρίζουν και τι κάνουν και οι μεγάλες εταιρείες όπως Facebook, Google κλπ. Εδώ ε, να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι και το κράτος οφείλει να είναι διαφανές όσον αφορά τις πληροφορίες τις οποίες πρέπει να δημοσιεύει, αλλά όταν ο πολίτης εμπιστεύεται τα δεδομένα του σε ιδιωτικές εταιρείες, οργανώσεις ή δεν ξέρω τι, αμέσως δημιουργείται μια σχέση. Και θα πρέπει τότε αυτός ο επεξεργαστής των δεδομένων να ανακοινώνει τι κάνει με τα συγκεκριμένα δεδομένα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, καλούνται τώρα οι ομιλητές να απαντήσουν. Να αρχίσουμε με τον κύριο Λεάντρη. Ας αρχίσουμε με την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ ασφαλώς θα χρειαστούμε περισσότερους ερευνητές. Είναι αλήθεια όμως ότι έχουμε και μεταξύ και από τη, τούτη την πλευρά του Ατλαντικού μερικούς από τους καλύτερους ερευνητές και μάλιστα και ορισμένους από αυτούς που έφτιαξαν τη τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια, σημαντικό είναι να μπορέσουμε να τους κρατήσουμε εδώ στις ευρωπαϊκές εταιρείες. Γι' αυτό χρειάζεται απλά να φτιάξουμε εταιρείε με ηθικές αξίες και θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε ερευνητές και επιστήμονες σε αυτές τις εταιρείε. Να τους δώσουμε δηλαδή τις δυνατότητες να κάνουν έρευνα και να εφαρμόσουν την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Αν είστε όπως εμείς εταιρεία μεγάλων μαζών δεδομένων, χρειάζεται να έχετε στη διάθεσή σας και σημαντικούς ερευνητές και να έχετε και την υποδομή, ώστε να μπορούν να ερευνούν για τεχνητή νοημοσύνη καθημερινά. Και να τους δώσετε και επαρκή ποσά δεδομένων για να μπορούν να κάνουν την έρευνα. Αυτό ακριβώ κάνουμε εμείς. Άλλοι βεβαίως πηγαίνουν κατευθείαν σε Google, Facebook κλπ. Αλλά στη Γαλλία για παράδειγμα, όταν το Facebook ξεκίνησε την ομάδα του τεχνητής νοημοσύνης, πήγε στη Γαλλία, διότι γνώριζε ότι εκεί υπάρχει, υπάρχει μεγάλος αριθμός ε, τέτοιων ερευνητών. Παίρνει 15 από αυτούς, φτιάχνει ένα κτίριο στο Παρίσι, τους βάζει εκεί και τώρα λέει ότι «Α ναι, κάνω τεχνητή νοημοσύνη». Απλώς έρχεται εδώ, παίρνει τους ανθρώπους δηλαδή, τους οποίους εμείς έχουμε εκπαιδεύσει και τους εντάσσει στο σύστημα αυτό αναλύσεων για να κάνουν ε, ανάλυση. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι όντως χρειάζεται να δαπανίσουμε πολλά στην παιδεία, στην εκπαίδευση, να βοηθήσουμε τους ερευνητές μας και τους μηχανικούς μας να μπορέσουν να εργαστούν με ένα μέγιστο αριθμό όγκο δεδομένων και με την καλύτερη δυνατή τεχνολογία. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Αλλά πέρα από αυτό πρέπει να τους δώσουμε την ικανότητα να ε, βασιστούν σε ευρωπαϊκές αξίες. Και αυτό το θέλουν πολύ Θέλουν να εργαστούν για επιχειρήσεις που έχουν και πιστεύουν σε αξίες, που έχουν ηθικές αξίες. Και ευρωπαϊκές αξίες είναι οι αξίες των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Δεν είναι τίποτα αμεληταίο όταν μιλούμε για αξίες ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και ο κανονισμό GDPR στην πραγματικότητα αυτό είναι. Βάζουμε δηλαδή, ε, ε, κάνουμε νόμο κάτι που μέχρι τώρα ήταν μια απλή δήλωση. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό τώρα στην Ευρώπη να αρχίσουμε να επενδύουμε σε εταιρείε οι οποίες εφαρμόζουν τους ευρωπαϊκούς νόμους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί χρειαζόμαστε να έχουμε την τελευταία λέξη τη τεχνολογία. Μην θεωρήσετε όμω ότι αν ρίξουμε όλα μα τα λεφτά στην εκπαίδευση θα φτάσει, ότι αυτό θα αρκέσει για να προσελκύσουμε όλους αυτούς τους σημαντικούς ερευνητές σε ευρωπαϊκές εταιρείες. Βεβαίως και χρειαζόμαστε την εκπαίδευση, βεβαίως και χρειαζόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά χρειάζεται να επενδύσουμε και στις εταιρείε μας από τη στιγμή που σέβονται τις αξίες. Αυτά για την εκπαίδευση. Ευχαριστώ να ε, δώσω το μικρόφωνο, αν με επιτρέπετε, στην ε, συνάδελφό μου για να απαντήσει για άλλα θέματα βιοτρικά δεδομένα κλπ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να απαντήσω στο δίλημα των φυλάκων που αναφέρετε κι εσείς. Ε, βεβαίως δεν λειτουργούμε σε κενό ως ερευνητές. Ε, ε λειτουργούμε ως ελεγκτές δεδομένων. Μας δεσμεύουν οι αρχές ιδιωτικότητας από το σχεδιασμό. Μας δεσμεύει το άρθρο 89 για συγκεκριμένες απαιτήσει για την έρευνα και θεωρώ πως αυτό το οποίο θα πρέπει να εφαρμόσουμε συνολικά και για την έρευνα της πληροφορικής είναι κάτι συγκρίσιμο με αυτό το οποίο υπάρχει στην ιατρική. Δηλαδή, μία υποχρεωτική εξέταση δεοντολογίας των μεγάλων ερευνητικών έργων. Αν θα θυμάστε, η Cambridge Analytica είχε πρόσβαση ως ερευνητής στα δεδομένα του Facebook και δεν ε, είχε σωστό έλεγχο. Εγώ θα ήθελα λοιπόν ένα συμβούλιο δεντολογίας που θα εξετάζει τα ερευνητικά μας έργα, θα μας δίνει το OK και τουλάχιστον για τα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα να υπάρχει κάποιο αρμόδιο για την προστασία των δεδομένων που θα συνεργάζεται μαζί μα και θα μα βοηθάει να εφαρμόζουμε ακριβώ την ιδιωτικότητα από τη φάση του σχεδιασμού. Και ε, αντιλαμβάνομαι, για να περάσω στην ερώτηση του Ισπανού εκπροσώπου, πως ε, οι απαιτήσει του κανονισμού μπορεί να είναι πολύ δυσκολότερες όταν μιλάμε για πρωτογενή έρευνα όπως ε, είναι συχνά στην ιατρική όπου υπάρχουν πολλά δεδομένα και οι ερευνητέ δεν ξέρουν τι ψάχνουν καν όσον αφορά τους διάφορους συσχετισμούς και νομίζω πω οι αρχές προστασίας δεδομένων πρέπει να κάτσουν μαζί με του ερευνητέ και να βρουν λύσει για τις δεοντολογικές ευθύνες και το πώς μπορούν οι αξίες του κανονισμού να μεταφραστούν στην πράξη για να είναι δυνατή και η έρευνα. Γιατί νομίζω ότι αξίζει και για την πρόοδο της κοινωνίας. Για να απαντήσω για το ίντερνετ των αντικειμένων. Για να είμαι σαφής το ίδιο θα ισχύει και για τα ιατρικά δεδομένα. Το ίντερνετ των αντικειμένων σημαίνει πως όλα τα δεδομένα που λαμβάνουμε από όλα τα αντικείμενα γύρω μας. Παραδείγματος χάρη δεν ξέρω αν ξέρετε την NetAtmo, την εταιρεία αυτή που πουλάει κάποιους ε, υγροποιητές ε, που έχετε στο σπίτι σας ε, και σας δίνουν επίσης κάποιες πληροφορίες για την κατάσταση της ατμόσφαιρας, την ρήπανση κτλ. Έχουν πουλήσει γύρω στο ένα εκατομμύριο κομμάτια σε ολόκληρο τον πλανήτη. Εάν είναι κάποιος συνδεδεμένος λοιπόν με τον ετάτμο μπορεί κάποιος να πει μπορεί να πει πως αυτός είναι ο καιρός εδώ και εκεί και παραπέρα και στον επόμενο δρόμο. Οπότε το σκεπτικό τώρα είναι ότι αν σκεφτούμε όλη αυτή τη συλλογή των δεδομένων υπάρχουν δύο τρόποι να συλλεχθούν. Πρώτον, έχουμε πρόσβαση σε όλες αυτές τις συσκευές, τους πελάτες, ποιος το έχει αγοράσει, ποια είναι η θερμοκρασία στο δωμάτιό του, στο σπίτι του, τι κάνει, είναι μέσα, έξω, είναι πιο ψηλή θερμοκρασία γιατί υπάρχει κάποια δραστηριότητα. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δούμε το τι κάνει ο άλλος μέσα στο σπίτι του. Ή ο δεύτερος τρόπος, σύμμορφο συμμορφούμενοι με την οδηγία, βλέπουμε ανώνυμα τα δεδομένα. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι σε διαμέρισμα ή όχι. Το μόνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι ο καιρός. Τι θερμοκρασία δείχνει το μηχάνημα. Και με βάση αυτό μπορούμε να προβλέψουμε τον καιρό εκεί, στο συγκεκριμένο δρόμο. Αυτό είναι σημαντικό για τους χρήστες, αλλά γιατί να έχουμε την πληροφορία το αν είναι το δικό στο μηχάνημα ή το δικό μου. Μπορούμε αυτό να το εφαρμόσουμε αναλογικά σε οτιδήποτε άλλο στο ίντερνετ των πραγμάτων. μπορεί να παίξουμε με την τεχνητή νοημοσύνη, με πολλά δεδομένα που να συλλέγουμε από όλο το ίντερνετ των αντικειμένων. Παραδείγματος χάρη στην Quant έχουμε υπογράψει με την A2A στην Ιταλία που παρέχει ηλεκτρισμό και υπηρεσίες και μας στέλνουν πληροφορίες, παραδείγματο χάρη, από το Μιλάνο και το τι γίνεται. Και έχουμε όλα τα δεδομένα. Εάν δεν ακολουθήσουμε τον κανονισμό, ξέρουμε αν είστε στο ποδήλατο ή στο τραμ ή στο μουσείο. Αλλά σκεφτείτε το ίδιο, αλλά χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι ποιος. Ξέρουμε τότε πού είναι τα ποδήλατα, αν θέλετε ένα ποδήλατο, ξέρουμε πού είναι το τραμ και αν έρχεται και αν μπορείτε να πάτε στο μουσείο επειδή είναι ανοιχτό. Αλλά χωρίς να είναι προσωπικά τα δεδομένα. Είναι λοιπόν σημαντικό να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα για το ίντερνετ των αντικειμένων που πρώτα απ' όλα θα έχει ανώνυμα τα δεδομένα και θα τα χρησιμοποιεί μετά για να δίνει στους ε, καταναλωτές ε, και στους Ευρωπαίους και σε ολόκληρο τον κόσμο, γιατί αυτό μπορεί να γίνει παντού, να ε, δώσουμε πραγματικές απαντήσεις, χωρίς να ξέρουμε αν χρησιμοποιώ το πράγμα εγώ ή εσύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να σκεφτούμε έτσι αυτήν την οδηγία, γιατί έτσι μπορούμε να παίξουμε με την τεχνητή νοημοσύνη χωρίς να υπάρχει η ανάγκη προσωπικών δεδομένων. Και για την υγεία, για, τα, για την βιοιατρική έρευνα, για τους ερευνητές. Είναι ακόμη χειρότερη Κατά έχω μία ερώτηση, αλλά θα, θα τα πω στα γαλλικά για να είμαι σαφής, μην κάνω κάποιο λάθος. Pour moi et pour et pour des... Για μένα και για όλους υπάρχει ένα θέμα. Το θέμα είναι, έχουμε μηχανικούς, έχουμε ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης και έχουμε και πλατφόρμες συλλογή δεδομένων και ικανότητες επεξεργασίας τους. Θεωρείτε ότι οι μηχανικοί μου είναι σε θέση να γνωρίζουν εάν το κύτταρο είναι καρκινογόνο ή όχι χωρίς να το εξετάσουν πρώτα οι γιατροί το τελικό αποτέλεσμα της ανάλυσης. Θα πρέπει λοιπόν να αναμίξουμε ερευνητές, γιατρούς, μηχανικούς, ειδικού τεχνητής νοημοσύνης. Να είμαστε ικανοί να τους βάλουμε όλους αυτούς σε μια πλατφόρμα την πλατφόρμα αυτή, να τη συνδέσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη που θα μας επιτρέψει να συσχετίσουμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κάπου αλληλοσυνδέονται, γιατί αυτό σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, και τελικώ η επιστροφή όλου αυτού να έρθει σε εμά και να φτάσει στους γιατρούς και στα νοσοκομεία. Να το πω ακόμα πιο ευθέω. Ποιο είναι το μέρο εκείνο του κόσμου που διαθέτει τα καλύτερα ιατρικά προσωπικά δεδομένα η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι. Η Γαλλία σήμερα, για παράδειγμα, γνωρίζω καλά τη χώρα αυτή, έτσι δεν είναι, έχει τα καλύτερα ποιοτικά ε, ιατρικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα. Και μόνο το γεγονός ότι θα μπορούσαμε να τα ανωνυμοποιήσουμε θα μας επέτρεπε να έλθουμε να σας προσφέρουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα τεχνητής νοημοσύνης εξυπηρετώντας τα νοσοκομεία, τους γιατρούς και τους ειδικούς μας. Δεν σας λέει κανεί, μάλλον δεν σα λέμε εμείς, ότι θα ζήσετε χίλια χρόνια αν πάτε να δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα στο Google. Εμεί λέμε να δώσουμε πράγματα σε αυτούς που γνωρίζουν. Κανένα δεν ζει ούτε και στη Silicon Valley, ούτε και μία μέρα πέρα από το θάνατό του. Και αυτά είναι, μιλούμε για σήμερα. συνδυασμό ανάμεσα στου ερευνητέ μα και στα ιατρικά δεδομένα ανωνυμοποιημένα που μπορούμε να τα διαθέσουμε, να τα διοχετεύσουμε σε πραγματικούς γιατρούς, σε πραγματικά νοσοκομεία, ώστε να εγγυηθούμε ότι τα δεδομένα σας δεν θα πουληθούν παραπέρα στην ασφαλιστική εταιρεία, στον Α, στον Β. Σε όλους μπορεί να βγάλουν κάποιο κέρδος από το αν εσείς αρρωστήσετε. Τα παιδιά, τα οποία μπορεί να γεννηθούν με μια αναπηρία, θα έχουν κάποιο μειονέκτημα στη ζωή, διότι η αναπηρία του θα είναι γνωστή στα προσωπικά του δεδομένα. Μπορούμε να φτιάξουμε λοιπόν σήμερα τεχνητή νοημοσύνη σε μαζικό επίπεδο, χωρί να γνωρίζει κανεί, έχω εγώ γρήπη, έχετε εσεί γρήπη, έχει ο τρίτο γρήπη. Είναι δυνατόν να γίνει. Σα παρακαλώ λοιπόν. Μην σπάσουμε την εφαρμογή του κανονισμού χώρα σε χώρα. Είναι τρόπος να προστατεύσουμε τον καταναλωτή και να επιταχύνουμε την χρήση των δεδομένων. Και κυρίως αυτό θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε την πρωτοπορία μας στα δεδομένα που διατηρούμε, σεβόμενοι τα δικαιώματα των ανθρώπων. You missed your calling as a politician. okay. Elections next year, right? No. Ready not. Depends what party. I shouldn't encourage you. Working next year. These, day, these days, the you, year never, after. you never know these days. Um, Δεν εκλογές χρόνο. Όχι, όχι, λέει κύριος Λέαντρη. Θα δουλεύω. Λοιπόν, μια που μιλήσατε τόσο πολύ και τόσο όγκλητα προέκυψαν άλλες δύο ερωτήσεις. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο κομμάτι για την ε, οδηγία για την αστυνομία. Ούτε ο Πολ Μπράιτπαρτ μίλησε. Λοιπόν, θα ακούσουμε τις ερωτήσεις ε, και μετά. Κύριος Μάρτιν ε, Τόλεντάνο και ο κύριος Φιντέλ από την Ισπανία και οι δύο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λογικά από τα όσα ακούσαμε προκύπτει το συμπέρασμα ότι είμαστε σε μια διαδικασία που πρέπει να ελέγξει πολύ σημαντικές ε, εξουσίες, δηλαδή εταιρείες που έχουν μια ένα μέγεθος, έναν όγκο μάλλον δεδομένων που τις τοποθετούν σε θέση ισχύω απέναντι στους πολίτες και στο, ε, ίδιο των κρατών στην Ευρώπη. Η ιστορία είναι η ιστορία της εξουσίας των κρατών. Περιορίσαμε τα κράτη που από το να μπορούν να έχουν στοιχεία στη διαθεσή τους που να μπορούν να βλάψουν τους πολίτες τους. Ε, τώρα όμως τα δεδομένα αυτά είναι στα χέρια εταιριών που έχουν εμπορικά συμφέροντα και που μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν και ενάντια στους πολίτες Συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν, όμως πιστεύω πως είναι σημαντικό να μπορούμε σε αυτή τη νομοθετική διαδικασία προσαρμογής του κανονισμού να έχουμε ένα μέσο το οποίο θα μπορεί να ε, χειριστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βλέπουμε πώς κάθε χώρα σταδιακά θα εγκρίνει την νομοθεσία του, για να δούμε δηλαδή πώς χρησιμοποιεί αυτό το μέσο, τι καινοτομίε έχει εισάγει, πώς νομοθέτησε και από το αρχικό σχέδιο, νομοσχέδιο μέχρι τη τελική έγκριση. Να έχουμε δηλαδή ε, έτσι ένα εργαλείο για αυτούς που δεν έχουν ακόμα νομοθετήσει και για να επαληθεύουμε κατά πόσο όντως αυτή η νομοθεσία οδηγεί στην εφαρμογή του κανονισμού. Όσον αφορά τα ιατρικά ζητήματα, να πω ότι ως άνθρωπος που υποφέρει από κάποια ασθένεια είμαι, ανησυχώ πάρα πολύ τα στοιχεία μου μπορεί να χρησιμοποιηθούν για μια έρευνα και γι' αυτό θα πρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες να έχουν τη δυνατότητα να προστατεύσουν τον ασθενή με ανωνυμία. Να υπάρχει δηλαδή ένα εργαλείο αποτελεσματικό και θα πρέπει αυτό να ισχύει για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, κυρία Πεντέχου. Εγώ θέλω να επανέλθω μισό λεπτό στο θέμα της βιοιατρικής και της έρευνας, της συγκατάθεσης και των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν για την ε, εξέλιξη εδώ. Η απέτηση εγκατάθεση ενός ενημερωμένου πολίτη είναι κάτι το απαρέκλειτο στην βιοιατρική γιατί μπορεί όμως αυτό να αποτελέσει εμπόδιο για την βιοιατρική έρευνα και συγκεκριμένα στην Ισπανία. Ο κανονισμός θέτει στα κράτη-μέλη και στην νομοθεσία τους ε, αυτό το ζήτημα και το σχέδιο δεν τροποποιεί την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά την έρευνα και για την υγεία που στη χώρα μου διέπεται από μία νομοθεσία του 2007 και από ε, ένα διάταγμα. Επιτρέπει έτσι πιο ευέλικτη νομοθεσία όσον αφορά την ε, ιατρική έρευνα Νομίζω πως αυτό αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τις ε, επιτροπές διοντολογίας όσον αφορά την έγκριση και τη διευκόλυνση της ε, ιατρικής έρευνας. Αυτό δεν περιλαμβάνεται ε, σε αυτές τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δεν συμφωνώ και πολύ με την κυρία Μπαρνάου που είπε ότι επειδή δεν ξέρουμε τι λύση θα δοθούν ε, σε αυτά τα προβλήματα που θα προκύψουν, ε, θα πρέπει να συνεδριάζουμε. Εμείς είμαστε φουλ μέσα στην νομοθετική διαδικασία. Κάνουμε αυτή τη δουλειά μας και εξετάζουμε τις τροπολογίες, να συνεδριάζουμε για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Για μας θεωρώ πως είναι ήδη εργά. Είμαστε υπέρ της ε, να, να φτιαχτεί μια νέα νομοθεσία μια νέα νομοθεσία που θα επιτρέπει στην πρακτική να δοθούν λύσεις σε αυτήν την ε, περίπτωση. Ο κ. Μπράικπαρτ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων για τις ερωτήσεις τους. Να ξεκινήσω με το θέμα της ιατρικής έρευνας, καθώς δεν είναι όμω ένα τομέα όπου κάνουμε πολλή δουλειά εμεί από την Νούμητη, όμω υπάρχουν κάποια. Ε, κάποιες σκέψεις που μπορούν να βοηθήσουν τόσο για το θέμα του πεδίου της έρευνας και του πεδίου της συγκατάθεσης, ε, τα εκτιμώντας, ε, ε, παρέχουν περιθώριο ελιγμού. Αντί να βιαστούμε λοιπόν για να στέξουμε νέα νομοθεσία, καλό θα ήταν, ε, προτείνω εγώ, να χρησιμοποιήσουμε αυτέ τι ιδεολογικέ σκέψει στι μέγιστε του δυνατότητε να ερμηνεύσουμε τι διατάξει του Γενικού Κανονισμού. Γιατί ειδικά για την ιατρική έρευνα ορίζεται ότι η συγκατάθεση δύναται να δίνεται με ευρύτερο τρόπο, χωρί ακριβώ να καταλαβαίνει κανεί τι σημαίνει η ιατρική αυτή έρευνα, γιατί είναι δύσκολο για τον ε, μη γιατρό να καταλάβει ακριβώς περί τίνος πρόκειται ή για ποιο λόγο θα χρησιμοποιηθούν ακριβώς τα δεδομένα του. Για την έρευνα λοιπόν πιστεύω πως υπάρχει περιθώριο ελεγμού μέσα στο κανονισμό από τη στιγμή που γίνεται με το σωστό τρόπο. Σωστό σημαίνει όσο, με όσο μεγαλύτερη διαφάνεια γίνεται αλλά και με δοντολογικό τρόπο να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα. Και εδώ συναντούμε δυσκολίες όταν έχουμε να κάνουμε με μεγαλύτερες εταιρείε που μπορεί να μην επεξεργάζονται τα δεδομένα με δεοντολογικό τρόπο ή να μην είναι απόλυτα δεοντολογικές στην προσεγγίση τους. Ακόμα και αν έχουν θεσπίσει ανεξάρτητα εποπτικά όργανα ή επιτροπές διοντολογίας. Επίσης, ε, όπως είδαμε πρόσφατα από έρευνες, διαπιστώνουμε πως υπάρχουν πολλές αρχές προστασίας δεδομένων και αποφάσει αυτών που δείχνουν ότι όσο μεγαλύτερος είναι κάποιο οργανισμός, τόσο μεγαλύτερη ευθύνη έχει για τη συμμόρφωση προς την νομοθεσία και να ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων τι σκοπεύει να κάνει. Η ευθύνη δηλαδή μεγαλώνει ανάλογα με την μέγεθο και τη εταιρεία. Τέλος, για την, για την παρακολούθηση των εθνικών νομοθεσιών που, αναφέρθηκαν οι Ισπανοί βουλευτές, είναι κάτι που κάνει ακριβώς η Νούμη ένα από τα ερευνητικά μας προγράμματα. Παρακολουθούμε όλες τις εθνικές εφαρμοστικές νομοθεσίες και τις μεταφράζουμε και τις δημοσιεύουμε στα αγγλικά από τη στιγμή που εγκρίνονται. Εμείς προσδοκούμε τη τελική εκδοχή της γαλλικής νομοθεσίας για να τη μεταφράσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Μάλιστα, σύντομες παρεμβάσεις παρακαλώ από την κυρία Μαρνάου και από τον κύριο Λεάνδρη. Πολύ σύντομη να είστε παρακαλώ για να περάσουμε στην επόμενη συνεδρία. συμφωνήσω με τον Πολ Μπράιτπαλτ ε, το να νομοθετούμε γρήγορα, ειδικά όσον αφορά την βιοιατρική έρευνα ε, είναι κάτι το οποίο θα είναι βεβαιασμένο. Εγώ θα ήθελα να δω πώς θα ερμηνεύσουν οι αρμόδιες ε, αρχές προστασίας δεδομένων τις απαιτήσει του κανονισμού, ειδικά για έρευνα μεγάλων δεδομένων και πρωτογενή έρευνα, στον βιοιατρικό τομέα και θα ήθελα να δω άλλες ε, λύσεις. Γιατί να βασίζεται η βιοιατρική έρευνα και στην συνένεση, αλλά και στα ανώνυμα δεδομένα, σε νέες τεχνολογίες όπως ε, η ιδιωτικότητα στην μάθηση της ε, τεχνητής ε, νοημοσύνης πριν ε, φτάσουμε να δούμε για το εάν μια ευρεία συνένεση επαρκεί για αυτό το πλαίσιο. Από την άποψη της, του κλάδου μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι μπορούμε να δουλέψουμε με ανώνυμα δεδομένα Υπάρχουν τρόποι να δουλέψει κανείς με τα ιατρικά δεδομένα με καθαρό τρόπο, με ιδεοντολογικό τρόπο και σεβόμενοι τον ε, γενικό κανονισμό. Τώρα, όταν επανέρχονται στο ε, νοσοκομείο, στον γιατρό σας, στα χέρια δηλαδή του ειδικού, εκείνος ξέρει ποιος είστε και θα μπορέσει τελικά να σας δώσει την καλύτερη θεραπεία, την καλύτερη αγωγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ομιλητές μας για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Περνάμε λοιπόν τώρα στο τελευταίο τμήμα. Στην αστυνομική δικαιοσύνη. Να έρθουν παρακαλώ οι ομιλητές εδώ πέρα. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό και ειδικά η δική μου πολιτική ομάδα πάλεψε για να παραμείνει εντός του κανονισμού τότε αυτό ακριβώς ε, μιλάμε για τους εναρμονισμένους ε, κανόνες ε, για την επεξεργασία δεδομένων από τις διοκτικές αρχές, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του νομοθετικού πακέτου. Και νομίζω ότι είναι επίτευγμα πραγματικά στο πλαίσιο των δύο νομοθετημάτων. Καλωσορίζουμε λοιπόν εδώ πέρα τον κύριο Κρίστιαν Βίζε Σβάνμπεργκ, ο οποίος είναι αρμόδιος λειτουργός για την ιδιωτικότητα και τμήματάρχης αρμόδιας μονάδα στην αστυνομία της Δανίας, τον κύριο Λιβιέ Μικόλ, τμήματάρχη τη Αρμόδια Μονάδα στην Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη τη Κομισιόν και την κυρία Μάγια Μόλτσικ, την Βρετανική Επιτροπή Προστασία. Με συγχωρείτε την Επιτροπή Προστασία Δεδομένων του Βερολίνου. Λοιπόν, ο κύριος Σβάνμπεργκ για 10 λεπτά. Σα ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. που με καλέσατε σήμερα να μιλήσω για τις πτυχές, ε, τις αστυνομικές της ε, σχετικής οδηγίας ήταν προαπαιτούμενο η Δανία να, για να μπορεί να έχει μια στενή σχέση με την Europol να εφαρμοστεί ο σχετικός νόμος πριν από την 1η Μαΐου 2017. Θα σας πω λοιπόν το τι κάνουμε στην Δανία με τη νέα αυτή οδηγία. Να σας πω βεβαίως πως δεν μπορώ εγώ να αναφερθώ σε πολιτικά ζητήματα και ζητήματα τα οποία αφορούν την ίδια την ε, οδηγία όταν ε, κοιτάμε το εάν έχει επιτευχθεί η σωστή ισορροπία όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τις διοκτικές αρχές. Και πριν προχωρήσω παρακάτω να σας πω ότι πριν ενταχθώ στην αστυνομία δούλευα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ε, στην αρχή προσωπικών δεδομένων και είχα και εγώ επί Προεδρίας της Δανίας στο Συμβουλίο Υπουργών εργαστεί για την σύνταξη αυτού του νομοθετικού πακέτου. Σήμερα λοιπόν είμαι υπεύθυνο της Μονάδας Προστασίας ε, δεδομένων. Έχουμε 11 άτομα στην μονάδα μας και είμαστε αυτοί οι οποίοι κοιτάμε το πώς η αστυνομία της Δανίας εφαρμόζει και συμμορφώνεται με τους κανόνες προστασίας δεδομένων. Εάν δούμε λοιπόν το ζήτημα αυτό, Νομίζω ότι μπορώ να πω ότι το προσωπικό το δικό μου είναι βεβαίως ενήμερο για τις ευθύνες που έχουν για την εφαρμογή των ε, κανόνων με τρόπο λογικό και αναλογικό. Και βεβαίως ε, πρέπει πάντα οι πληροφορίες ε, που προκύπτουν από τι έρευνες να παραμένουν πάντα εμπιστευτικές ε, και φυσικό είναι να θέλουμε και να προστατεύσουμε την αστυνομία να έχει τη δυνατότητα να κάνει την δουλειά της και να τηρούμε ταυτόχρονα την εμπιστευτικότητα και την προστασία της ακαιρεότητας των δεδομένων και βεβαίω ε, και οι αστυνομικοί θέλουν να συμμορφώνονται με τον νόμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, οι νέε απαιτήσει ε, δεν είναι μια αλλαγή την οποία αισθανόμαστε. Έχουμε λοιπόν κάποιες υποχρεώσεις, έχουμε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα, παραδείγματο χάρη το δικαίωμα που έχουν τα άτομα να ενημερώνονται για το ότι τα δεδομένα τους ε, τηρούνται. Είναι κάτι το οποίο είχαμε βεβαίως ήδη ως διαδικασία από τον, την οδηγία του 1995 αλλά είναι μια καινοτομία όσον αφορά τις διοκτικές αρχές. Ε, τώρα μπορούμε να πούμε ότι σαφώς πρέπει να ενημερώνονται οι πολίτες. Εν ολίγης είναι δύσκολο να γίνει μια έρευνα για ένα έγκλημα αν ενημερώνουμε ε, κάποιον ότι ε, είναι υπό έρευνα. Οπότε ίσως θα χρειαστεί να υπάρξει μια καθυστέρηση σε αυτή την ενημέρωση. Και βεβαίως κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια είναι το πότε ακριβώς θα πρέπει να γίνεται αυτή η ενημέρωση. Στην Δανία Προσπαθούμε ακριβώς να δούμε το πώς η αστυνομία γενικώ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα. Το αναφέρουμε στην ιστοσελίδα μας. Υπάρχουν αφήσει στα αστυνομικά τμήματα. Εξηγούμε δηλαδή στους πολίτες ε, το, τι διαδικασίες υπάρχουν και πόσο μπορούν αν θέλουν να υποβάλουν κάποια καταγγελία να προσφύγουν για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και ακριβώς αυτό είναι το θέμα της επεξεργασίας των μαζικών δεδομένων όπως και η υπόλοιπη κοινωνία έτσι και οι αστυνομικές αρχές έχουν μεγάλες προκλήσεις στο πλαίσιο αυτό έχουμε τις εμπειρίες που έχουμε ε, και στο Europol και βλέπουμε ότι η αποτελεσματική χρήση των δεδομένων είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις που έχει και η κοινωνία. Η χρήση όμως των ε, μαζικών δεδομένων σημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις και από την αστυνομία και από αυτούς οι οποίοι μας παρέχουν τα μέσα, τα εργαλεία για να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες αυτές. Η αστυνομική οδηγία λοιπόν είχε κάποια θετικά αποτελέσματα γιατί τώρα ο νόμος απαιτεί από την αστυνομία της Δανίας να διασφαλίσει ότι συμμορφώνεται με τους κανόνες προστασίας δεδομένων, κάτι το οποίο βεβαίω μας διευκολύνει και μας όταν ζητάμε κάτι από τους προμηθευτές μας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για το τι αποτελέσματα είχαν οι κανόνες αυτές κανόνε αυτοί με για την αστυνόμευση στην πράξη. Να αναφερθώ δηλαδή στο πώς καθορίζουμε ποιοι κανόνες ισχύουν σε ποιες περιπτώσεις, γιατί όταν μιλάμε για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Συνεργασία. ήταν δύσκολο, παραδείγματο χάρη, να, να κρίνουμε το εάν οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων ε, θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με αυτήν την οδηγία ή με κάποια άλλη οδηγία. Έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια συγκεκριμένη ερμηνεία των κανόνων, να γνωρίζουμε γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα και να δούμε για ποιον σκοπό μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν οι αρχές που εμπλέκονται. Οπότε μια λύση θα μπορούσε να είναι ότι οι αστυνομικές ε, και άλλες αρχές και οι αρμόδιες αρχές για την προστασία των δεδομένων να καθίσουν μαζί να δουν ποια θα μπορούσε να είναι μια πρακτική απάντηση με διαφάνεια σε αυτό το ζήτημα. Έτσι θα είναι ευκολότερο και για τις αρχές και για τους πολίτες. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μωραές, ελπίζω τα, παράδειγμα, τα παραδείγματα αυτά να είναι χρήσιμα στην Επιτροπή σας και είμαι βεβαίως στην διάθεσή σας και για ερωτήσεις ακόμα και τεχνικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα περνάμε λοιπόν στον κύριο Ολιβιέ Μικόλ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Βασικά θα ήθελα στην αρχική μου εισήγηση να καλύψω τρία στοιχεία. Πρώτον, ας πούμε, τα, τα κύρια στοιχεία αυτής της νέας νομοθεσίας που κάποιες φορές τα παραμελούμε και περισσότερο ε, εστιάζουμε το γενικό κανονισμό. Ε, επίσης κάποια σημαντικά ζητήματα δεν θα, δεν διατρέξω όλα τα άρθρα βεβαίω, αλλά θα τονίσω κάποια σημαντικά ζητήματα που περιλαμβάνονται στην οδηγία και έπειτα να πω, κάνουμε μια, έναν απολογισμό για το πού βρισκόμαστε τώρα γιατί η επίσημη προθεσμία για τη μεταγραφή της νομοθεσίας ήταν η 6η Μαΐου. Ποια είναι τα βασικά κεντρικά στοιχεία. Αυτή η οδηγία αποτελεί τμήμα του εις δέσμης προστασία δεδομένων μαζί με τον Γενικό Κανονισμό. Ε, η προθεσμία για τη μεταγραφή, όπως σας είπα, είναι η 6η Μαΐου, ήταν η 6η Μαΐου και πρακτικά θα έπρεπε να είναι η 25η Μαΐου μαζί με τον Γενικό Κανονισμό και βλέπουμε ότι για πολλά κράτη-μέλη αυτή είναι η ημερομηνία στην οποία στοχεύουν γιατί βλέπουν τις δύο αυτές νομοθεσίες ως δέσμοι. Αυτή η οδηγία αντικαθιστά την απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου του 2008. Περνάμε δηλαδή από ένα μέσο του τρίτου πυλώνα σε οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Δηλαδή πρόκειται για μια λισαβονοποίηση των κανόνων. στόχοι, κύριοι στόχοι είναι κοινοί, δηλαδή υψηλό επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο της ε, αστυνομικής συνεργασίας και της ποινική δικαιοσύνης, καθώς και ε, η δημιουργία μιας ομαλότερης ε, ροής ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τέλος συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών αδικημάτων εγκλημάτων στην Ευρώπη. Η κυρία αλλαγή είναι ότι καλύπτει τόσο την ε, χώρια όσο και την διασυνοριακή ε, κατάσταση. Έχουμε ισχυρότερα δικαιώματα για ένα υποκείμενο δεδομένων. Έχουμε εμπνευστεί από το Γενικό Κανονισμό το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα για διόρθωση, διαγραφή ή οτιδήποτε άλλο. Και έχουμε ένα πολύ σημαντικό σημείο που είναι η άμεση πρόσβαση ε, του υποκειμένου δεδομένου στα δικαιώματά του. Τι σημαίνει η άμεση πρόσβαση, ότι ένας πολίτης μπορεί να πάει κατευθείαν στην αρχή και μόνο αν τα δικαιώματα αυτά περιορίζονται θα έπρεπε να περάσει από την αρχή προστασίας δεδομένων το υποκείμενο. Η άμεση πρόσβαση είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι κάτι που δεν είχαμε με βάση την προηγούμενη απόφαση πλαίσιο. Επίσης εισάγεται νέα αρχή παρόμοια με του γενικού κανονισμού δηλαδή ε, προστασία δεδομένων από το σχεδιασμό ή εξορισμού, συμπεριλαμβάνεται η ε, λογοδοσία των ίδιων των αρχών, για παράδειγμα για την ε, διεξαγωγή αξιολόγησης κινδύνου. Επίσης πρέπει να ορίσουν αρμόδιο υπεύθυνο ε, κοινοποίηση των ρήξεων των δεδομένων, παραβιάσεων των δεδομένων, όπως στον Γενικό Κανονισμό και υποχρέωση για ε, διατήρηση ε, ημερολογίων είναι ίσως αυτή η πιο δύσκολη πρόκληση για πολλές από τις αρχές γιατί, γιατί έχει αντίκτυπο στο σύστημα πληροφορικής τους. Όσον αφορά τις διεθνείς μεταφορές, ε, η προτιμόμενος διεύλος είναι επίσημο έτοιμα από τις αρμόδιες αρχές, αλλά έχουμε επίσης τη δυνατότητα άμεσης συνεργασίας από τους παρόχους των υπηρεσιών υπό συγκεκριμένους όρους. Αυτά πολύ συνοπτικά είναι τα κεντρικά στοιχεία. Αλλά να τονίσω και κάποια συγκεκριμένα σημαντικά ζητήματα που έχουμε εντοπίσει στο πλαίσιο της συζήτησης με τα κρατημέλη. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, κάτι που ανέφερε και ο κ. Βάνμπεργκ μόλις, η οδηγία η ισχύει για τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη δίωξη. Δεν ισχύει ας πούμε, για τις αρχές που διευκολύνουν ε, καθήκοντα επιβολής του νόμου και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την οριοθέτηση ε, ανάμεσα στην οδηγία ε, της αστυνόμευση και την οδηγία, τον γενικό κανονισμό δίνεται τη δυνατότητα στα κρατημέλη να έχουν την ίδια αρχή προστασίας δεδομένων για τις δύο ε, νομοθεσίες και αυτό είναι πολύ θετικό το, το γεγονός ότι τα περισσότερα κρατημέλη επέλεξαν να έχουν κοινή αρχή προστασίας δεδομένων και για το γενικό κανονισμό και για την οδηγία περί αστυνόμευσης. Μόνο το Βέλγιο έκανε διαφορετική επιλογή. και ε, ε, έτσι θα υπάρχει περισσότερη συνοχή ανάμεσα στο Γενικό Κανονισμό και την Οδηγία περί αστυνόμευσης. Όπως αναφέραμε, ε, πρόκειται για τεχνικά ζητήματα, τα οποία όμως είναι δύσκολο να εφαρμοστούν όταν υπάρχουν ήδη συστήματα πληροφορικής και πρέπει να αλλάξει αρχιτεκτονική για να μπορείς να παρακολουθείς τα δεδομένα. Και γι' αυτό και υπάρχει και μια πρόβλεψη για μακρύτερη μεταβατική περίοδο μέχρι το 2023 και ίσως και το 2026 σε εξαιρετικές περιστάσεις. Και βλέπουμε ότι πολλά κράτη-μέλη όπου τώρα φτιάχνουν το σύστημα είναι ευκολότερο να το εφαρμόσουν από την πρώτη μέρα, ενώ οι υπόλοιποι θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν τη μακρύτερη αυτή μεταβατική περίοδο. Αυτό που επίσης είναι σημαντικό είναι το ζήτημα του ποιος εποπτεύει το δικαστήριο. Γιατί η οδηγία αυτή ορίζει ότι η εποπτική αρχή δεν είναι τα εποπτικά δικαστήρια και άλλη ανεξάρτητη δικαστική αρχή. Και τότε το ερώτημα τίθεται ποια είναι αυτή η άλλη ανεξάρτητη δικαστική αρχή. Ο ίδιος εισαγγελέα που έχει το ίδιο επίπεδο ανεξαρτησίας όπως και ο δικαστής. Και αυτό υπάρχει στην Ιταλία, αλλά όχι σε όλα τα κράτη-μέλη, διότι οι εισαγγελίε δεν είναι απαραίτητο πλήρω ανεξάρτητοι. Τώρα, οι εξουσίε οι αρμοδιότητε τη προ... Ε, αρχής προστασίας των δεδομένων είναι πιο μικρή από ότι αυτή που προβλέπει το γενικό κανονισμό, όμως πρέπει να είναι αποτελεσματική και πρακτική, δηλαδή ερευνά, συμβουλεύει στην πράξη και αυτό που βλέπουμε είναι ότι πολλά κράτη-μέλη αποφάσισαν τελικά να δώσουν το ίδιο επίπεδο αρμοδιοτήτων στην ε, αρχή προστασίας δεδομένων και στην αρχή ε, για την οδηγία περί Εναρμονίζουν δηλαδή τις αρμοδιότητες των αρχών προστασίας δεδομένων και για τις δύο νομοθεσίες. Σημαντικό είναι ότι υπάρχει άμεση πρόσβαση από το υποκείμενο των δεδομένων στις αρχές, σε ορισμένα κράτη-μέλη. Η ισχύουσα πρακτική λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει. Υπάρχει βεβαίως δυνατότητα να περιοριστούν τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων υπό την οδηγία περί αστυνόμευσης, όπως πούμε το δικαίωμα στην ενημέρωση κτλ. Αλλά ε, αυτό ε, θα πρέπει να ερμηνευθεί με περιορισμένο τρόπο. Δεν μπορούμε να έχουμε δηλαδή μια, έναν γενικό περιορισμό για όλα τα υποκείμενα δεδομένων. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω κάποιες διαφορές με τον γενικό κανονισμό. Όπως γνωρίζετε, και αυτό έχει τονιστεί και παλιότερα, έχουμε ε, ε, ε, συγκεκριμένη νομική βάση, έξι νομικές βάσεις για την προστασία δεδομένων, ενώ για την αστυνομία έχουμε μόνο μία, δηλαδή τον νόμο. Δεν υπάρχει άλλη αρχή διαφάνειας στην οδηγία αυτή, αν και υπάρχει αρχή της δίκαιης δίκης, που σημαίνει επίσης κάποιο βαθμό διαφάνειας. Η έννοια του περιορισμού των δεδομένων ισχύει επίσης και εδώ, γιατί μιλάμε για δεδομένα τα οποία δεν πρέπει να είναι υπερβολικά. Δεν λέει ότι περιορίζονται στα αυστηρός απαραίτητα. Δίνεται δηλαδή λίγο μεγαλύτερη ευελιξία στις αστυνομικές αρχές. τα δεδομένα πρέπει να ε, σβηστούν ή περιοδικώς πρέπει κανείς να εξετάζει αν χρειάζεται να διατηρήσει τα στοιχεία. Και αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα που συνδέεται με την ειδική, το ειδικό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής. Πού βρισκόμαστε, έχω λίγο, λιγότερο από ένα λεπτό, πού βρισκόμαστε μετά από τη διετή μεταβατική περίοδο στην Κομισιόν, όπως και με το Γενικό Κανονισμό, έχουμε εκτεταμένες πολυάριθμες ε, συνεδριάσεις με τις εθνικές αρχές ώστε να προετοιμάσουμε την εφαρμογή της δέσμης προστασίας δεδομένων, δηλαδή ε, την οδηγία περί και τον γενικό κανονισμό και καλωσορίζουμε τη γνωμοδότηση της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 που δίνει πολύ ενδιαφέρουσες, ε, ενδιαφέροντα στοιχεία για διάφορα περιπτώσεις, για διάφορα θέματα όπως ας πούμε ποιο είναι το χρονικό όριο για τη διατήρηση των στοιχείων, το θέμα της εγγραφής στο ημερολόγιο, και ένα σωρό άλλα χρήσιμα ε, ζητήματα είναι πολύ χρήσιμη γνωμοδότηση μπορεί να καθοδηγήσει τις αρμόδιες αρχές. Πού βρισκόμαστε τώρα λοιπόν. Κατάσταση πρόοδο, όπως είπα, τα περισσότερα κρατημέλη, τα μισά μάλλον θα έλεγα, θα έχουν το ίδιο μέσο για μεταγραφή της οδηγίας επιβολής του νόμου και για την εφαρμογή του γενικού κανονισμού του Γενικού Κανονισμού. Μόνο τρία κράτη-μέλη έχουν κοινοποιήσει μέχρι στιγμής, Γερμανία, Σλοβακία και Λιθουανία. Και βασικά, εάν συνοψίσουμε χονδρικά έχουμε 7 κράτη-μέλη που πάνω κάτω είναι στην, εντός των προθεσμιών του Μαΐου. Ορισμένα 7 είναι κάπως πίσω, δηλαδή προβλέπουν τον Ιούνιο και την εβδομάδα μετά και μετά άλλα μισά κρατημέλη που δεν είναι ξεκάθαρο γιατί είναι ακόμα στην κοινοβουλευτική διαδικασία το θέμα. Σε κρατημέλη, κάποια κρατημέλη υπήρξαν εκλογές, οπότε έχει καθυστερήσει η διαδικασία. Αυτά λοιπόν για την ώρα και βεβαίως υποστηρίζουμε, εφόσον είμαστε εδώ, πολλοί εκπρόσωποι είστε εδώ από τα Εθνικά Κοινοβουλία, υποστηρίζουμε και σας παροτρένουμε να επιταχύνετε στο δικό σας επίπεδο την υιοθεσία των απαραίτητων ε, νομοθεσιών για την μεταγραφή της οδηγίας για την επιβολή του νόμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να με συγχωρείτε γιατί χρειάστηκε να λείψω για λίγα λεπτά. Η κυρία Σμόλτσικ. Δέκα λεπτά παρακαλώ, όχι περισσότερο. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, και από μένα ευχαριστίες που μου επιτρέπετε σήμερα να σας απευθύνω τον λόγο. Εν ώψη των νομοθετικών δραστηριοτήτων στο εθνικό επίπεδο θεωρώ σημαντικό στην ευρωπαϊκή, στο ευρωπαϊκό επίπεδο να παρακολουθείτε ακριβώς η δραστηριότητα των Εθνικών Βουλών για τη μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο, διότι υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευθεί ο στόχος της εναρμόνισης στο ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω και της υπερβολικής χρήσης των ρητρών ανοίγματο. Ως επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων του Ομόσπονδου Κρατηδίου Βερολίνου μπορώ να σε εξηγήσω μόνο τι συμβαίνει παροιμήν. Γνωρίζω όμως ότι τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι άλλες γερμανικές αρχές προστασίας δεδομένων. Έως τώρα στο Βερολίνο η οδηγία Εσωτερικών και Δικαιοσύνης δεν έχει ακόμα μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. Αποφάσισε λοιπόν η Βουλή του Βερολίνου να συνδυάσει την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και των δύο, οδηγίας και κανονισμού. Το σχέδιο της νέας νομοθεσίας για το Βερολίνο πάντοτε βρίσκεται σε κοινοβουλευτική συζήτηση και θα εγκριθεί πριν από τις θερινές διακοπές. Πρόκειται για νόμο που θα περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις που ισχύουν για τις δημόσιες αρχές στον χώρο του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας Εσωτερικών και Δικαιοσύνης. Μόνο σε συγκεκριμένα ε, σημεία ε, θα υπάρχουν ειδικοί νόμοι, όπως για παράδειγμα για τις αρχές επιβολής του νόμου. Ωστόσο είναι προβληματικό ότι η δική μου αρχή παρόλες τις κατ' επανάληψη δεν έχει λάβει τη δυνατότητα να υποβάλει εισηγήσει σχετικά για παράδειγμα με την αστυνομική νομοθεσία και να λάβει γνώση των σχεδίων. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο κατά την δική μας εμπειρία δεν επιτρέπει να γνωρίζουμε, να έχουμε επαρκή τεχνογνωσία για το τι πρόκειται να συμβεί. Τώρα, πότε θα υποβληθούν τα σχετικά σχέδια στην Βουλή του Βερολίνου δεν είναι γνωστό. Την Τετάρτη της προηγούμενης εβδομάδας τέθηκε υπόψη μου το σχέδιο του νέου νόμου για την ε, προστασία των δεδομένων. Και μόλις μια μισή μέρα μετά, δηλαδή εχθές, έγινε η ακρόαση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής του Βερολίνου. Ήταν τόσο σύντομο το διάστημα που δεν μπορέσαμε να εξετάσουμε το σχέδιο νόμου σε όλες τις λεπτομέρειες. Με μια σύντομη ματιά πάντως διαπιστώσαμε τα εξή προβλήματα. Τα ήθελα μάλιστα να τα θέσω υπόψη σας. Άρθρο 47, παράγραφος 2 της Οδηγίας Εσωτερικών και Δικαιοσύνης. Εμείς ως Αρχή Προστασίας Δεδομένων πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα την αρμοδιότητα προσφυγής. Αυτό όμως μπορεί να έχει αποτελέσματα μόνο εάν είναι δεσμευτική για τους υπευθύνου και επομένως νομικά εκτελεστή. Στο σχέδιο ωστόσο νόμου δεν περιλαμβάνονται αυτές οι διατάξεις. Αντιθέτως, για το πεδίο εφαρμογή της Οδηγίας Εσωτερικών και Δικαιοσύνης εξακολουθούν να μιλούν για τα ατελή μέσα της διαπίστωσης ελλείψεων και της αμφισβήτησης. Αυτά τα μέτρα μπορούν να τα απαιτήσουν οι ε, αρμόδιες αρχές, αλλά είναι μη δεσμευτικά. Στο παρελθόν το διαπιστώσαμε αυτό δυστυχώς πολλές, σε πολλές περιπτώσεις και έχουμε μακρού χρόνου εμπειρία με την χρήση των νομικών αυτών μέσων, τα οποία δεν λήφθηκαν υπόψη από τις αρμόδιες αρχές όταν τα προωθήσαμε εμείς. Είχαμε ζητήσει λοιπόν συγκεκριμένες διατάξεις στο νέο νόμο. Η πρότασή μας ήταν να υιοθετηθούν και από το νόμο του Βερολίνου τα άρθρα 47 παράγραφος 2 της Οδηγίας ε, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, πρόταση όμως η οποία δεν έγινε δεκτή. Ακόμα χειρότερα, επιμένουν στις παλές ρυθμίσεις με, την, ε, με ούτε καν αιτιολόγηση και δεν μιλούν καθόλου για τις ε, νέες ευρωπαϊκές διατάξεις. Αν παραμείνουν οι ρυθμίσεις αυτές ως έχουν, τότε η αρχή μου δεν θα έχει τις αναγκαίες αρμοδιότητες που προκύπτουν από το άρθρο 46 παράγραφος 1 υποπαράγραφος α, δηλαδή εποπτεία και παρακολούθηση των διατάξεων που εκδίδονται δυνάμει της οδηγίας. Το πρόβλημα αυτό υπάρχει και στον τομέα της ομοσπονδιακής νομοθεσίας στην οποία βασίστηκε και ο νομοθέτης του Βερολίνου. Πρόκειται για ανεπαρκείς ρυθμίσεις και μάλιστα ακατανόητες, διότι θα έπρεπε να είναι δεσμευτικές και επομένως να εξετάζονται και από τα δικαστήρια. Υπάρχει και άλλη μια δυσχέρεια στο νέο νόμο, ότι δεν προβλέπονται δηλαδή ρυθμίσεις για την εκτέλεση. Ακόμα και αν ο Βερολινέζος νομοθέτης παραχωρήσει στην αρχή μου αρμοδιότητες για την έκδοση εντολών, αυτές δεν θα μπορούν να εκτελεστούν αναγκαστικά, διότι δεν υπάρχουν οι αναγκαίες νομοθετικές διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση. Και αυτό αφορά και την οδηγία αλλά και τον κανονισμό. Και στους δύο τομείς, σύμφωνα με τον νομικό σχεδιασμό που γίνεται έως τώρα, δεν προβλέπεται αναγκαστική εκτέλεση. Κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει μέγας κίνδυνος για την εφαρμογή των ε, ευρωπαϊκών ρυθμίσεων. Και εμεί αυτή την κριτική την έχουμε ασκήσει κατ' επανάληψη. Τώρα, σύμφωνα με το άρθρο 57 της οδηγίας, υπάρχει καθήκον του εθνικού νομοθέτη να προβλέψει κυρώσει στην περίπτωση παραβιάσεων, καθώς και να δώσει και συγκεκριμένους ορισμούς των μέτρων που λαμβάνονται. Αυτά όμως έχουν μεταφερθεί ε, ανεπαρκώς στο εθνικό δίκαιο. Εμείς ζητήσαμε να προβλέπονται και χρηματικές ποινές διότι οι χρηματικές ποινές ιδίω ιδίως παραβιάσεις μικρότερης ε, βαρύτητας είναι αποτελεσματικές κυρώσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα ατομικές παραβιάσεις έγινε δεκτή αυτή η πρόταση. Δεν προβλέπονται όμως κυρώσεις για παραβιάσεις των διατάξεων για την προστασία δεδομένων από project μέτρα των υπεύθυνων αρχών. Αυτό ισχύει επαναλαμβάνω, και για το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία και για το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Περιλήφθηκε επίση στο νομοσχέδιο τη ε, ε, Βερολινέζικη Βουλή κάτι το οποίο, έχει, ε, το οποίο είναι αμφισβητούμενο σε ό,τι αφορά δηλαδή τον αντίκτυπο των παραβιάσεων. Είναι δυνατόν σύμφωνα με τη νέα διάταξη, παρόλο που συνεχίζει να εξετάζεται η υπόθεση και πριν να λήξουν οι προθεσμίες, να αρχίσει η εργασία εφόσον, λέει ο νόμος, είναι, είναι ε, κατεπήγον το θέμα. Βέβαια, πρόκειται για έννοιες οι οποίες μπορούν να ερμηνευθούν με διαφορετικό τρόπο. Αλλά δεν εξασφαλίζεται η προστασία δεδομένων και επιτρέπεται να γίνουν κάποιες ενέργειες πριν να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την αρχή προστασίας δεδομένων. Ούτως ή άλλως βεβαίως η προθεσμία είναι υπερβολικά σύντομη και στον ψηφιοποιημένο κόσμο είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί το αποτέλεσμα οποιασδήποτε παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. Στον τομέα της διαφάνειας και των ε, δικαιωμάτων των θυγωμένων, ο νομοθέτης και για την εφαρμογή της οδηγίας, αλλά και για την προσαρμογή στον κανονισμό, δεν εξαντλεί τα περιθώρια περιορισμών, αλλά τα υπερβαίνει κιόλας. για να μπορέσει να παίξει διορθωτικό ρόλο η αρχή μου, αυτό δεν επιτρέπεται σε πολλά σημεία. Σύμφωνα με το υφιστάμενο σχέδιο υπάρχουν τομείς όπου τα φυγόμενα πρόσεπα... δεν λαμβάνουν ενημέρωση, ούτε μπορούν να ζητήσουν οι σχετικέ πληροφορίε να διατεθούν σε μένα, επικεφαλή τη Αρχή Προστασία Δεδομένων. Θα υπάρξουν λοιπόν περιπτώσει όπου το σημαντικότερο δικαίωμα του θυγωμένου, δηλαδή η ενημέρωσή του, δεν πληρούνται. Και αυτό σημαίνει ότι υπονομεύονται σημαντικέ λειτουργίε ελέγχου. Και κάτι ακόμα, το οποίο δεν αφορά μονάχα τη δική μου αρχή προστασία δεδομένων, αλλά νομίζω όλε τι γερμανικέ αρχέ προστασία δεδομένων, γνωρίζετε όλοι ότι η εφαρμογή και της οδηγίας και του κανονισμού θέτουν πολύ περίπλοκα ζητήματα και προβλέπουν πολλές νέες υποχρεώσεις για τις αρχές προστασίας δεδομένων. Υπάρχει επίσης ανάγκη, ζήτηση δηλαδή, και από την οικονομία και από άλλες ε, κρατικές αρχές. Γι' αυτό προβλέπει και η οδηγία και ο κανονισμός ότι κάθε αρχή προστασίας δεδομένων εξοπλίζεται στελεχώνεται και εξοπλίζεται με όλα τα αναγκαία μέσα για να μπορέσει να εκτελέσει αποτελεσματικά τα θήκοντά της. Πολλές, ωστόσο, αρχές προστασίας δεδομένων απέχουν πολύ. Πολλές έχουν πολύ ανεπαρκές ε, προσωπικό και στελέχωση. Δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη ο ρόλος τους και παρόλες τις ε, αιτήσει που έχουμε υποβάλει δεν λαμβάνονται υπόψη. για το Βερολίνο μπορώ να πω ότι εμείς έχουμε ένα ε, προσωπικό ενθουσιωδών ε, συνεργατών οι οποίοι αναμένουν να μπορέσουν να εργαστούν για την εφαρμογή του νέου κανονισμού. Αναμένουμε να είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το επόμενο ε, χρονικό διάστημα και θα συνεργαστούμε ευχαρίστως με τους άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους μας. Το αν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις με την εφαρμογή των διατάξεων των αρχών μάλλον το, τις οδηγίες και του κανονισμού με τόσο περιορισμένο στελεχικό δυναμικό, εμένα αυτό με απασχολεί πολύ. Θα πρέπει να έχει κανείς διαρκώς υπόψη του ότι εάν δεν είναι δυνατόν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους με αντικειμενικά ικανοποιητικό τρόπο, τα στελέχη αυτό, αυτά θα χάσουν οποιοδήποτε ενθουσιασμό και αυτό θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο διότι θεωρώ ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Προχωρούμε σε ένα ψηφιακό μέλλον και ο μόνος τρόπος για να προστατευτεί το άτομο είναι αυτός. Θα χαρώ πολύ να συνοδεύσει κριτικά το ευρωπαϊκό επίπεδο της προσπάθειές μας και θα ήθελα να ε, ολοκληρώσω με τα λόγια αυτά και να σας ευχαριστήσω πολύ για την προσοχή σας. Και περνάμε τώρα κατευθείαν στι ερωτήσεις και παρεμβάσεις βουλευτών από τα Εθνικά Κοινοβούλιο. Πρώτα κυρία Κοζοπολίου την Ελλάδα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση επισήμανση στον κύριο Κριστιαν Βίζε ε, ε, Σβάνμπερκ, γιατί ακούμπησε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα, δηλαδή τη χρυσή τομή ανάμεσα στην προστασία των δεδομένων και την, ε, και την ασφάλεια για τις έρευνες που διεξάγει η αστυνομία για το έγκλημα το εθνικό ή το διασυνοριακό Θέλω λοιπόν, εδώ ο κανονισμό έχει προβλέψει την τήρηση δύο αρχών, τη αναλογικότητα και τη αναλαχιστοποίηση. Ξέρετε τι σημαίνουν αυτά, να μην τα αναλύω. Θέλω μόνο να ρωτήσω αν στην πράξη αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και αν υπάρχει κάποια πρακτική που ε, είναι χρήσιμο να την ε, μεταφέρετε εδώ. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλησπέρα σας. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, μιλώντας για προσωπικά δεδομένα, μπορούμε να μιλήσουμε φαινός για ανθρώπινα δικαιώματα και από την άλλη βεβαίως έχουμε την αστυνομία και την χρήση της τεχνολογίας και πάντα ακριβώς προκύπτει αυτό το ζήτημα της θεμελιώδους δυσπιστίας που υπάρχει απέναντι στην αστυνομία. Σε κάποιες από τις χώρες μας είχαμε κάποιες αρνητικές εμπειρίες. Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα είναι το εξής η ε, ανείχνευση του κυβερνοεγκλήματος, ε, το οποίο δεν έχει σύνορα. Ανεξαρτήτως του πόσο προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να διορθώσει την κατάσταση μέσω κανονισμών, οι κλιματικές οργανώσεις είναι πάντα ένα βήμα μπροστά και πάντα θα βρουν έναν τόπο που θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν ανενόχλητες. Το άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι το θέμα των προσόντων των διοκτικών αρχών, το θέμα του εξοπλισμού τους και το θέμα της τελέχωσης. Αυτά οπωσδήποτε είναι ζητήματα πάρα πολύ ε, σημαντικά. Ε, όταν μιλάμε επίσης για το κυβερνοέγκλημα, ένα κομμάτι αυτού είναι και η κλοπή προσωπικών δεδομένων ε, και διαρρήξεις μέσα σε η κλοπή καρτών και εικονικές θα λέγαμε διαρρήξεις ε, της ιδιωτικότητας. Μπορούμε λοιπόν εδώ πέρα να ορίσουμε εμείς κανόνες ε, και νόμους, αλλά είναι δύσκολο να βρεθεί το όριο μεταξύ της ιδιωτικότητας ε, και των μεγάλων συμφερόντων. Ξέρουμε πλέον ότι οι πληροφορίες είναι ένα εμπορεύσιμο αγαθό. Και αυτό σημαίνει ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο Ε, αποτελούν, ε, θα έλεγα, κάτι ανάλογο με τα κρυπτονομίσματα. Και όταν μιλάμε και για τις ε, πληροφορίες και τις αστυνομικές αρχές και τις ποινικέ κυρώσεις, το θέμα είναι και ο έλεγχος επί των αστυνομικών και δικαστικών αρχών και μετά έχουμε το θέμα της αποθήκευσης αυτών των δεδομένων και πάλι προκύπτει το ερώτημα του ποιος είναι ο υπεύθυνος, ποια θα είναι η περίοδος διακράτησης αυτών των δεδομένων, ποιος θα τα αποθηκεύσει και ποιος θα ασκεί έλεγχο. Κάποιες χώρες, όπως ακούσατε, προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα. Αλλά Αναμένουμε βεβαίω ε, και τις προτάσεις της Κομισιόν. Αν κάθε κράτο μέλο ε, προσπαθεί να βρει τον δρόμο με τις ε, δικές του υπηρεσίες, αυτό θα σημαίνει ότι κάποια κράτη-μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίσουν επιθέσεις. Έχουμε δει ήδη τέτοιες επιθέσεις όταν εκλάπησαν δεδομένα από εταιρείε και άρχισαν τότε τα κράτη-μέλη να αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό είναι το θέμα. Τα αυτά και εμένα. Θα... έχουμε δύο γύρους ε, ερωτήσεων. Θα ακούσουμε τις ερωτήσεις, μετά τις απαντήσεις των ομιλητών. Ε, όποιοι θέλουν να πάρουν το λόγο ε, μπορούν να το ζητήσουν και μετά θα ακούσουμε τις απαντήσεις των εισηγητών μας. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Εντάξει, άλλος κανείς θέλει να πάρει το λόγο. Δεν θα υπάρξει δεύτερος γύρος, μόνο ένας γύρος. Εντάξει. Ωραία, λοιπόν, και παρακαλώ να είστε σύντομοι. Κύριος Σβόνη, από το Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω πολωνικά. Po Σας ευχαριστώ πολύ για τη διοργάνωση της σημερινής συνεδρίασης. Εγώ εδώ και πολλούς μήνες ζητούσα τη διοργάνωση ε, μιας τέτοιας συνεδρίασης ε, σε σχέση με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού. Η σημερινή ε, συνεδρίαση δείχνει ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα αλλά και πολλές ευκαιρίες. Επίσης ε, δείχνει ότι είμαστε έτοιμοι να, ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δείξουμε εμπιστοσύνη και να αξιοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα ερμηνευτούν ε, οι διατάξεις του νέου κανονισμού. Η ισχύς των εθνικών ε, θεσμών που θα ερμηνεύσουν στου ε, στους κανονισμούς θα στηρίξουν τους πολίτες αλλά και τον επιχειρηματικό κόσμο στην εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων. Πολλοί ομιλητές είπαν ότι δεν υπάρχει πουθενά ετοιμότητα 100% σε κανένα από τα κρατημέλη και αυτό είναι πολύ ισχυρό μήνυμα. Υπογραμμίστηκε δε από πολλούς από τους ομιλητές ότι πολλά από τα προβλήματα που σχετίζονται με την προώθηση των όσων προσφέρει η οδηγία και ο κανονισμός δεν είναι γνωστό. Δεν είναι γνωστά. Πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουν τι προτείνεται και πώς ισορροπείται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων με την εκτέλεση των διαφέρων καθηκόντων των διαφόρων αρχών που επίσης είναι για την ασφάλειά τους. Δεν υπάρχει ευκαιρία για μια επισκόπηση της κατάστασης στα διάφορα κράτη-μέλη όσον αφορά την πρόσβαση στη ε, προσωπικά δεδομένα άνευ περιορισμών ή όσον αφορά τους κανόνες που ορίζει αυτή η οδηγία όταν λέμε πως χρειάζεται να έχουμε έναν κατάλογο για ποινικά δικήματα, μιλάμε για γνωμοδότηση του δικαστήριου πριν ληφθεί η απόφαση. Σε ορισμένες χώρες όμως το δικαστήριο απλώς ενημερώνεται ε, ex post, όταν δηλαδή έχει χορηγηθεί πρόσβαση στα δεδομένα και σε κάποια κατημέρια δεν υπάρχει κατάλογος σοβαρών αδικημάτων. Όλα τα δικήματα εξετάζονται σαν να είναι σοβαρά δικήματα. Τίνουμε λοιπόν να εστιάζουμε στον κεντρικό γενικό κανονισμό. Αν δούμε όμως τα δικαιώματα των πολιτών, είναι σημαντικό να εξηγήσουμε αυτές τις λεπτομέρειες όσον αφορά τα θέματα αστυνόμευση, στο πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα δικαιώματά μας και οι αρχές επιβολής της νομοθεσίας θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης ποιοι είναι οι κανόνες στους οποίους πρέπει να υπακούν. Παρακαλώ να είστε σύντομος. Ο κύριος Σαμπατόσκας από την Λιθουανία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Οι συγητέ και οι συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια σήμερα υπογράμμισαν κάποιες πτυχές της οδηγίας και του κανονισμού τα δύο αυτά νομοθετήματα ορίζουν όρους και προϋποθέσεις για την επεξεργασία δεδομένων. Ωστόσο, έχουμε εδώ να αντιμετωπίσουμε ένα δίλημα ανάμεσα στην επιβολή του νόμου και των αρμοδίων αρχών, τις δραστηριότητε τους και τις, των κακόβουλων ε, ε, φορέων που μπορεί να είναι εγκληματίες ή άλλοι που θέλουν να βλάψουν τα προσωπικά δεδομένα. Ε, ορίζονται βέβαια ε, όροι και προϋποθέσεις για την πρόσβαση σε δεδομένα σε περιπτώσεις ε, πληροφόρησης για εγκληματίες, για πρόληψη εγκλημάτων, για συγκεκριμένα είδη εγκλημάτων. Υπάρχουν και εθνικές νομοθεσίες που ορίζουν τους κανόνες για τη συγκέντρωση των στοιχείων. Όμως, κάποιες φορές δεν αρκούν για τον εντοπισμό των εγκληματικών δραστηριοτήτων και τα στοιχεία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βρεθούν οι δράστες. Οπότε η ερώτησή μου είναι η Για πόσο καιρό μπορούν να αποθηκευτούν τα δεδομένα. Μια άλλη πτυχή που θέλω να αναφέρω είναι η τρομοκρατία, τα εγκλήματα τρομοκρατίας. Οι τεχνολογίες της ανοίγουν νέους δρόμους και νέες ευκαιρίες. Είμαστε σε θέση να έχουμε πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες για εγκλήματα που διοργανώνονται ή για τα ε, ε, ανθρώπους που αναμεγνύονται. Αυτό μπορούμε να το έχουμε άμεσα τη σημερινή ημέρα. Πιστεύετε ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα ισορροπίας ανάμεσα στην ε, πληροφορία που πρέπει να αποθηκευτεί και την πληροφορία που πρέπει να καταστραφεί. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν στοιχεία που είναι σημαντικά για τον εντοπισμό ενός εγκληματία αλλά τα δεδομένα αυτά μπορούν ήδη να καταστραφούν διότι το έγκλημα στο οποίο έχει προβεί αυτός ο άνθρωπος να καταστραφούν επειδή το έγκλημα έχει γίνει πολύ καιρό πριν. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Ο κ. Σούλερ από τη Γερμανία. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, διακόπτη ο πρόεδρος. Παρακαλώ ο προηγούμενος ομιλητής να κλείσει το μικρόφωνο του. Είναι δύο μικρόφωνα ανοιχτά και προκαλούν σύγχυση. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν, έλεγα κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τα μέλη του πάνελ για τις πολλές λεπτομέρειες που μας έθεσαν υπόψη. Πράγματι, υπάρχει ένα πλήθος πληροφοριών σχετικά με τον βασικό κανονισμό και είναι σημαντικό να προβάλλονται και να μεταφέρονται και στις πολλές συζητήσεις που γίνονται με, τις, ε, τους πολίτες. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξή. Πώς μετρούν οι αρχές προστασίας δεδομένων, ποια είναι η ατζέντα που έχουν, εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με τον κανονισμό. Κάνουν κάποια ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πεδίο αρμοδιοτήτων που διαθέτουν. διότι κυκλοφορεί εσφαλμένα η εντύπωση ότι οι αρχές προστασίας δεδομένων δεν περιμένουν τίποτε άλλο παρά να έχουν τη χαρά να δυσκολεύσουν τη ζωή των ανθρώπων, είτε πρόκειται για επιχειρηματίες, είτε πρόκειται για ε, χρήστες κλπ. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω αν γίνεται επικοινωνία προς τα έξω, προς το κοινό δηλαδή, και αν γίνεται και επικοινωνία των αρχών προστασίας δεδομένων και μεταξύ τους. Διότι αυτό είναι σημαντικό για να κινητοποιήσουμε και την κοινή γνώμη να αντιληφθεί περισσότερο και καλύτερα ποια είναι τα δεδομένα της προστασίας, ε, ποια είναι μάλλον ποιες είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες θα γίνει η προστασία δεδομένων. Θα είμαι σύντομο, λέει ο κ. Λόπε Αγγιλάρ. Έχω μιλήσει και στα προηγούμενα πάνελ. Έχω ερώτηση προς τον κύριο Νικόλ για τη, της Γενικής δικαιοσύνη, Δικαιοσύνης ό,τι αφορά το επίπεδο ετοιμότητα που διαθέτουν οι χώρε μέλη και σε ό,τι αφορά την διαθεσιμότητα και την δυνατότητα να εφαρμόσουν αμέσως την οδηγία η οποία αποκαλείται μεν πολύ directive δηλαδή ε, οδηγία αστυνομία, αλλά δεν περιλαμβάνει μονάχα την συνεργασία των αρχών επιβολής ε, του νόμου αλλά και για παράδειγμα του εισαγγελείς σχετικά με την προστασία της προσωπικής σφαίρας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και όχι μόνο στην εθνική νομοθεσία αλλά και σε ό,τι αφορά και την διαμεθοριακή συνεργασία διότι είδαμε τα τελευταία χρόνια μια επιδίνωση της διάθεσης ή μια μείωση της διάθεσης συνεργασίας των αρχών δικαιοσύνης και των εισαγγελικών αρχών μεταξύ των χωρών μελών της Ένωσης που έχει οδηγήσει σε επιδίνωση της δυνατότητας επίτευξης των στόχων των σχετικών νομοθετημάτων. Θα ήθελα να μάθω από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης σχετικά με την διάθεση εφαρμογής. Διότι πρόκειται για μια οδηγία, πολύ στερεκτή δηλαδή, η οποία ήδη έχει τεθεί σε ισχύ. Ήδη από τις 6 Μαΐου ενώ αναμένουμε την εφαρμογή του κανονισμού, η οδηγία ήδη εφαρμόζεται. Αυτό το πολύ directive είναι στην πραγματικότητα μια συντομία, μια συντομογραφία που δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται. Όταν λέγαμε απλώ οδηγία, κανεί δεν γνώριζε για ποια μιλούσαμε. Ήταν πραγματικά ανώνυμη. Άρχισαν λοιπόν να την αποκαλούν η αστυνομική οδηγία. Και όλοι ξαφνικά ανησύχησαν ή αγανάκτησαν ή τέλος πάντων άρχισαν να ενθουσιάζονται, αναλόγω με το σε ποιο τμήμα του πολιτικού φάσματος βρίσκεται ο καθένα, και ιδίω κάποιοι οι υπουργοί βέβαια στο Συμβούλιο Παρχών που δεν του πολύ άρεσε, με συγχωρείτε πολύ εσεί τα εθνικά κοινοβούλια, δεν γνώριζαν ε, δηλαδή όταν άκουγαν πολύ στα Ερέκτιβ τι είναι, διότι δεν ήθελαν καν να, να βάλει χέρι στι δικέ του αστυνομίε. Όχι, πρόκειται για ένα είδο συντομογραφία, γι' αυτό αρχίσαμε να την αποκαλούμε έτσι. Δεν είναι στην πραγματικότητα. Ε, συγγνώμη για την παρέμβασή μου αυτή. Η κυρία Στέβενς. Και μετά θα ακούσουμε τις ε, απαντήσεις από το πάνελ. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι ως στην Επιτροπή περί τρομοκρατίας αντιλαμβάνομαι ότι η τρομοκρατία και το ξέπλυμα χρήματο είναι παγκόσμια φαινόμενα που πρέπει να αντιμετωπιστούν παγκοσμίω. Το οικονομικό έγκλημα δεν σέβεται σύνορα και βεβαίω οι διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικές ε, λίστες υψηλού κινδύνου. Οπότε ο ιδιωτικό τομέα παίζει σημαντικό ρόλο στο να ε, βοηθήσει τα κράτη να σηκώσουν αυτό το βάρος. Και βεβαίως ε, ο κανονισμός ε, δεν ξέρω αν θα βοηθήσει ή όχι τον ιδιωτικό τομέα στο, στην δουλειά του, αλλά ίσως επηρεάσει το πώς, υπάρχει, το πώς γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων των ατόμων. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια αμφισημία στο άρθρο 23 όσον αφορά το δημόσιο συμφέρον. Θεωρώ ότι εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια για να υπάρχει ένα αποτελεσματικό καθεστώς καταπολέμησης του ξεβλήματο ε, χρήματος ε, και της ε, τρομοκρατίας. Σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε νομίζω με τις ερωτήσεις. Μπορούμε να επιστρέψουμε στους ομιλητές μας. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κύριο Σβάνμπεργκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να απαντήσω την ερώτηση της Ελληνίδας βουλευτού για την εμπειρία που έχουμε από την συλλογή μαζικών ε, δεδομένων. Να σας πω ξεκάθαρα πως ε, υπάρχουν ε, κάποιες προκλήσεις που αφορούν και το ότι τα πληροφορικά μας συστήματα είναι κάπως πεπαλαιωμένα και είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε τα ανέστηματα τα οποία θα είναι εξ αρχής προορισμένα για αυτήν την δουλειά και να σας πω και ειλικρινά είναι ζήτημα χρημάτων. Έχουμε... Αν έχουμε δηλαδή επαρκείς πόρους ε, για τα συστήματα αυτά τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν μεγάλους όγκους δεδομένων. Είναι μια πρακτική ε, πρόκληση, αλλά θεωρώ ότι είναι και φυσικό κομμάτι των δυνατοτήτων που έχουν οι αρχές να χρησιμοποιούν μαζικά δεδομένα, ε, πάντα οπωσδήποτε με λογοδοσία και θα πρέπει να είμαστε σε θέση να επιδείξουμε το πώς επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα. Ελπίζω να σας απάντησα. Να περάσω τώρα στον κύριο Μικόλ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις οι οποίες ήταν πολλές. Θα τις ομαδοποιήσω. Λοιπόν, υπήρχαν αρκετές ερωτήσεις ε, για τους πόρους, ε, για τις αρχές προστασίας δεδομένων και πράγματι είναι μια υποχρέωση του Γενικού Κανονισμού και της Οδηγίας τα κράτη-μέλη να δίνουν στις αρμόδιες αρχές ε, τους απαραίτητους ε, πόρους, ε, υλικούς και οικονομικούς. Αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο τόνισε η Κομισιόν στην ανακοίνωση του Ιανουαρίου που μας ε, πέρασε και είναι κάτι το οποίο επαναξιολογήσαμε και σήμερα στην ε, ανακοίνωσή μας ε, προς την ε, Σύνοδο Κορυφής όπου λέμε ότι ο Γενικό Κανονισμός είναι ένα βασικό στοιχείο και θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να έχουν τους απαραίτητους πόρους. Και από την άλλη υπάρχει ε, ανάγκη να έχουν ουσιαστικές αρμοδιότητες. Όταν τα κράτη-μέλη μεταφέρουν την οδηγία στην ομοθεσία τους πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα έχουν τις αρμοδιότητες οι αρχές προστασίας δεδομένων. Η οδηγία περί αστυνομίας έχει πιο γενικές διατυπώσεις γιατί ο γενικός κανονισμός καθορίζει τις αρμοδιότητες και το καθήκον και είναι κανονισμός και ισχύει απευθείας και βεβαίως ε, οι αρχές ε, έχουν ε, και τις ε, ιδιοκτικές αρχές, έχουν και τις δυνατότητες ε, της επιβολής. Και βεβαίως η οδηγία πρέπει να είναι αποτελεσματική, πρέπει να μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία. Για τους πόρους επίσης αξίζει να σημειώσουμε πως επαφίεται μεν στον εθνικό νομοθέτη να διασφαλίσει, στι εθνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι, αλλά βεβαίως και εμείς δίνουμε κάποιες επιχορηγήσεις στις αρχές προστασίας δεδομένων για να έρθουν σε επαφή με τους πολίτες, ειδικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Είχαμε δημοσιεύσει μια προκήρυξη η οποία ε, έχει κλείσει και κοιτάμε τώρα τις αιτήσει που λάβαμε. Επίσης υπάρχει το ζήτημα του πώς ε, θα ερμηνευτούν οι διατάξεις ε, και του κανονισμού και της οδηγίας. Και εδώ πέρα θα ήθελα να επισημάνω την δουλειά που έχει κάνει η ομάδα εργασίας του άρθρου 9 και υπάρχουν ήδη 10 κατευθυντήριες γραμμές που έχουν δημοσιευτεί, αφορούν ε, την οδηγία, τον κανονισμό αλλά και την αστυνομική οδηγία και όπως σας είπα αφορούν ε, συγκεκριμένα την ε, αστυνομική οδηγία. Και εδώ πέρα κοιτάω συγκεκριμένα το ερώτημα που έγινε το για πόσο καιρό θα πρέπει να διακρατούνται τα δεδομένα. Αν δείτε λοιπόν την γνωμοδότηση της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 δεν υπάρχει μια σαφής απάντηση που να λέει χι αριθμό ετών γιατί αυτό εξαρτάται από την φύση των δεδομένων αλλά υπάρχει ήδη στην ε, γνωμοδότηση αυτή μια πολύ χρήσιμη αρχή που ορίζει την αρχή της αναγκαιότητας, ε, δηλαδή να διατηρούνται τα δεδομένα μέχρι να επιτευχθεί ο σκοπός ε, και μόνο πρέπει να υπάρξει κάποια διάκριση μεταξύ των δεδομένων ενός υπόπτου, ενός μάρτυρα, υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες και να υπάρξει και μία αναλογή αντιμετώπιση, οπότε στην ε, γνωμοδότηση αυτή που προετοίμασαν οι αρχές προστασίας δεδομένων υπάρχουν διάφορες ε, απαντήσεις. Υπήρχε και μία ερώτηση για την ανακοίνωση που σχετίζεται περισσότερο με τον γενικό κανονισμό παρά με την αστυνομική οδηγία. Εδώ πέρα θα ήθελα να επισημάνω τα διάφορα εγχειρίδια, κατευθυντήριες γραμμές ε, κτλ. Τα οποία δημοσίευσε η Επιτροπή, ε, μεταξύ των οποίων 60 ερωταποκρίσεις για τα βασικά στοιχεία του κανονισμού σε όλες τις γλώσσες. Ε, έχουμε και εγχειρίδια ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους πολίτες. Και οπωσδήποτε ε, στο εθνικό επίπεδο οι εθνικές αρχές ε, θα διαδώσουν τις πληροφορίες αυτές στους πολίτες, στους ενδιαφερόμενους, αλλά προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε αυτή την βοήθεια μέσω αυτού του υλικού. Επίσης ετέθη το συγκεκριμένο ζήτημα της ετοιμότητας των κρατών μελών όσον αφορά την αστυνομική οδηγία ε, το ανέφερα αυτό και στην αρχική μου τοποθέτηση. Η κατάσταση ε, σωστά αναφέρεται ε, ότι η προθεσμία για μεταφορά ήταν η έκτημα ή Σε πολλές περιπτώσεις τα κράτη-μέλη έχουν το ίδιο μέσο αυτό για να εφαρμόσουν την ε, οδηγία και να υπάρξει και η προετοιμασία για τον κανονισμό. Για πολλά κρατημέλη λοιπόν θα είναι 21η Μαΐου. Αυτό το οποίο βλέπουμε αυτήν την στιγμή είναι ότι χοντρικά θα έλεγα τα μισά κράτη-μέλη θα ε, το έχουν κάνει εγκαίρως είτε α, ε, λίγες εβδομάδες μετά αλλά έχουμε και τα άλλα μισά κρατημέλη που θα καθυστερήσουν περισσότερο από μερικές εβδομάδες εάν δεν επιταχύνουν την ε, διαδικασία. Και θα ήθελα να παρακαλέσω πάλι τους βουλευτές ε, που είναι στην να επιταχύνουν την διαδικασία γιατί όπως λέτε το γεγονός ότι δεν είναι έτοιμα όλα τα κρατημέλη σημαίνει ότι θα υπάρχει ένας κατακαιρματισμός ε, του τοπίου προστασίας δεδομένων και είναι σημαντικό να είμαστε όλοι στο ίδιο σημείο οι αρχές προστασίας δεδομένων να έχουν τις απαραίτητες αρμοδιότητες και τους πόρους για να υπάρχει μια εφαρμογή, ε, αν όχι από την πρώτη μέρα, ε, τουλάχιστον τις επόμενες, σε ένα εύλογο διάστημα. Η κυρία Σμόλτσικ, ευχαριστώ και εγώ για τις ερωτήσεις, κυρίως σχετικά κατά πόσον οι αρχές προστασίας δεδομένων επικοινωνούν μεταξύ τους και κατά πόσο κάνουν και μια επικοινωνία προς τα έξω σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ε, οδηγίας. Στην πραγματικότητα έχουμε πάρα πολύ στενή ανταλλαγή απόψεων, όχι μόνο στο εθνικό επίπεδο, Βεβαίω η Γερμανία ω ομόσπονδα δομημένη χώρα έχει και την ε, ιδιαίτερη πρόκληση να αντιμετωπίσει των ε, διαφορετικών ενδεχομένω εφαρμογών ε, ή ερμηνεών που γίνονται στις διάφορες ε, διάφορα ομοσπονδα κρατήδια, αλλά και στην Ευρώπη υπάρχει πάρα πολύ έντονη ανταλλαγή απόψεων για να γίνει προσπάθεια να εξασφαλιστεί ότι οι κυρώσεις που προβλέπει ο οργανισμός αλλά και η οδηγία εσωτερικών και δικαιοσύνης να εφαρμόζονται ή δυνατόν με τον πιο ομοιογενή τρόπο. Δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, διότι αλλιώ δεν θα επιτύχουμε τον στόχο τη εναρμονίσεω και αυτό είναι σαφέ. Παρά τον ανεξάρτητο χαρακτήρα παραδοσιακά των αρχών ε, προστασία δεδομένων, τον οποίο ε, διαφυλάσσουν ω κόρηνο οφθαλμού. Για το ερώτημα κατά πόσον ε, το παρουσιάζουμε, το μεταφέρουμε αυτό και στην κοινή γνώμη, κάνουμε προσπάθεια. Κάνουμε προσπάθεια εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε βέβαια μέχρι τον τελευταίο. Εξαρτώμεθα και από τη συνεργασία των επαγγελματικών οργανώσεων, των ε, αντιπροσωπευτικών οργανώσεων, να μεταφέρουν δηλαδή και στις τάξεις των μελών τους το μήνυμα αυτό. Προσπαθούμε όμως να αντιταχθούμε σε αυτό τον πανικό που αρχίζει και εξαπλώνεται σιγά σιγά. Προσπαθούμε να αντιταχθούμε σε αυτό το κύμα ανησυχίας, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται στις 26 Μαΐου να αρχίσουμε αμέσως να επιβάλλουμε κυρώσεις, χρηματικά πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ή έστω και δεκάδων εκατομμυρίων, ότι βεβαίως θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή πάρα πολλών κριτηρίων ε, το πόσο σοβαρή ή βαριά θα κριθεί η παραβίαση σε κάθε περίπτωση και βεβαίως πάντοτε με απόλυτο σεβασμό των διατάξεων του κανονισμού και της οδηγίας εάν πρόκειται για μικρές παραβιάσεις, δεν θα οδηγηθούμε καν σε επιβολή κυρώσεων. Θα κάνουμε πρώτα, ε, θα εκδώσουμε πρώτα προειδοποιήσεις. Προσπαθούμε λοιπόν εντατικά και μέσω διαβουλεύσεων με ενδιαφερομένους φορείς να εξηγήσουμε ποια θα είναι η στάση μας, διότι για μας δεν έχει απολύτως κανένα νόημα να υποδαβλίζουμε την ανησυχία αυτή. Αυτό προσπαθούμε εμείς να εξηγήσουμε. Είναι ότι είναι πραγματικά κάτι σημαντικό, κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι εγκρίθηκε στο ευρωπαϊκό επίπεδο ο κανονισμός για να γίνει αντιληπτή η προστασία δεδομένων ως δικαίωμα των πολιτών που έχει μια θεμελιώδη σημασία και που ήταν αποτέλεσμα ενός κοπιώδους αγώνα και που είναι σημαντικό δικαίωμα να διατηρηθεί μέσα σε αυτόν τον όλο και πιο ψηφιακό κόσμο. Προσπαθούμε λοιπόν να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα. Από την άλλη μεριά οι ερωτήσεις δείχνουν ότι είναι και μια δύσκολη πορεία για τις αρχές προστασίας δεδομένων, γιατί από την άλλη μεριά είμαστε και υποχρεωμένες να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που προσφέρει ο κανονισμός, ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και τον στόχο της εναρμόνισης. Αν δεν υπάρχει απειλή των κυρώσεων δηλαδή, αυτός ο ανθρώπινος άλλωστε πειρασμός να καταστρατηγηθεί το πνεύμα του νόμου θα συνεχιστεί δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στην περίπτωση αυτή. Γι' αυτό χρειάζεται η απειλή των κυρώσεων και βεβαίω εν αμφιβολία θα επιβληθούν κιόλα. Αλλά όπω είπα, όπως είπα, όχι βέβαια στι πιο μικρέ παραβιάσει. Το ερώτημα τώρα σχετικά με την επιλογή. Είπα προηγουμένω ότι οι αρχέ προστασία δεδομένων είναι ανεπαρκώ τελεχωμένε και είναι αυτονόητο ότι δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να αξιολογήσουμε με την ίδια ένταση και την ίδια προσπάθεια όλες τις υποθέσεις που θα τεθούν υπόψη μας. Θα είμαστε υποχρεωμένες να βάλουμε κάποια κριτήρια, κάποια ιεράρχηση σχετικά με τις υποθέσεις που θα επιλέξουμε να ασχοληθούμε με αυτές. Βεβαίω πρωτίστως θα εκτελέσουμε τα καθήκοντα που μας επιβάλλει δεσμευτικά ο κανονισμός και η οδηγία κατά τα λοιπά, οι δραστηριότητες που θα αναλάβουμε εξαρτώνται βεβαίως από τα στοιχεία που θα τεθούν υπόψη μας. Θα αναγκαστούμε να κάνουμε κάποια αξιολόγηση της βαρύτητας των υποθέσεων. Θα δούμε πρώτα, θα προσπαθήσουμε να επιληθούμε πρώτα των πιο σημαντικών προβλημάτων. Βεβαίως, δειγματοληπτικά θα ασχοληθούμε και με άλλες υποθέσεις για να υπάρχει, να δημιουργηθεί ένας σεβασμός για την ε, τήρηση των διατάξεων. Κάποιος μίλησε προηγουμένως για την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις αστυνομικές αρχές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες την πραγματικότητα οι διοικητικές αρχές και ο συνολικός δημόσιος τομέας. Αυτό, η δυσπιστία αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο εάν συνεχιστούν οι προσπάθειες διαφάνειας και αν λάβουν σοβαρά οι αρχές αυτές η υπόψη της διατάξης του, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, διότι μόνο άνθρωποι οι οποίοι είναι ενημερωμένοι για το τι γίνεται στο δημόσιο τομέα με τα προσωπικά τους δεδομένα μπορούν να αποκαταστήσουν και την εμπιστοσύνη τους, γνωρίζοντας δηλαδή ότι δεν πρόκειται να παραβιαστούν τα δικαιώματά τους. Με τις ρήτρε ανοίγματο αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται και από τις αναγκαίες αντισταθμίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Οδηγούμαστε σιγά σιγά στο πέρας ε, των εργασιών μας. Ευχαριστώ πολύ τα μέλη των Εθνικών Βουλών για την ε, παρουσία σας στη διάρκεια των συζητήσεων και για τις ε, πολύ υψηλού επίπεδου παρεμβάσεις σας. θα λάβετε και το πρακτικό της ε, σημερινής συνεδριάσεως και νομίζω ότι με τη συζήτηση που κάναμε ανταποκριθήκαμε στο υψηλό επίπεδο της ε, διαβούλευσης. Ευχαριστώ βεβαίως και τους συναδέλφους μου ευρωβουλευτές, μέλη της Επιτροπής ε, Θεμελιωδών Ελευθεριών, δύο μεν μόνο. Ευχαριστώ όμως πάλι όλος ιδιαίτερος τους εθνικούς βουλευτές και με μεγάλη χαρά θα παρακαλέσω τον κύριο Ράλο Λομπάρτε του Ισπανικού Κοινοβουλίου να κάνει τις τελικές παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ και πάλι όλες και όλους. Έχει το λόγο κύριε. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχάς ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και την Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ για την ε, ευτυχή αυτή η πρωτοβουλία να διοργανώσει αυτήν ε, την συνεδρία ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Εντός 10 ημερών στις 25 Μαΐου θα αρχίσει μια νέα φάση στην ιστορία των προστασία δεδομένων στην Ευρώπη και θα ολοκληρωθεί μια διαδικασία που δεν ήταν μόνο μια διαδικασία των δύο τελευταίων ετών από τότε δηλαδή που εγκρίθηκε ο κανονισμός, αλλά μια διαδικασία των τελευταίων πέντε τουλάχιστον ετών από τότε δηλαδή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2012 υπέβαλε τις ε, προτάσεις ε, νομοθετικής πρωτοβουλίας για οδηγία και κανονισμό. Στις 25 Μαΐου λοιπόν θα ολοκληρωθεί μια διαδικασία που ε, χρονολογείται εδώ και 23 χρόνια όταν εγκρίθηκε η πρώτη οδηγία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων το 1995. Αυτό που ισχύει είναι ότι είναι βέβαιο πως σύντομα ε, διαπιστώθηκαν αδυναμίες και νέες προκλήσεις που είχαν να κάνουν με την ανάδυση νέων τεχνολογιών, με την έλλειψη εναρμόνισης ε, των ευρωπαϊκών κανόνων, με την δύσκολη και αναγκαία προσαρμογή των νομοθετικών κανόνων στις διεθνείς κανόνας μεταφοράς στοιχείων, δεδομένων και αναζήτηση συνοχής. Αυτή η πραγματικότητα μάλιστα δεν μπορούμε να ξεχνάμε, ότι πρέπει να ξεχάσουμε ότι παράλληλα Ακολούθησαν και νομικές και συνταγματικές αλλαγές ε, και συγκεκριμένα αναφέρομαι το 2000 ε, εγκρίθηκε ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά αναγνωρίστηκε ως ε, δικαίωμα θεμελιώδες η προστασία των προσωπικών δεδομένων και μετά η συνθήκη της Λισαβόνας που κατέστησε αυτό το χάρτη αναπόσταστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ε, νομοθεσίας. Όλα αυτά δεν είναι ξένα προς την εξέλιξη και προς το βήμα που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να παρουσιάσει τότε το σχέδιο κανονισμού και οδηγίας το 2012 που κατέληξαν μετά από τρία χρόνια στην έγκριση του κανονισμού και της οδηγίας μετά από μια μακρά συζήτηση, έντονη και τεταμένη συζήτηση κάποιες φορές που προκλήθηκαν από το φαινόμενο που το είδε και ο, που μας το θύμισε ο τότε πρόεδρος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και που έχει γραφτεί στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν υπήρχαν πολλές ε, ε, εμπειρίες τέτοιας πίεσης από τους λομπίστες ε, όπως είδαμε με αυτή το, τη δέσμη προστασίας των δεδομένων που σημαίνει ένα άλμα ποιοτικό φοβερό υπέρβαση των αδυναμιών του παλαιού νομικού πλαισίου μέσω της ε, ε, εξέλιξης αυτού του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, το άρθρο 8 και ε, οδηγία και απόφαση πλαίσιο που ίσχυαν τότε στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας και βέβαια ο κανονισμός αντικαθιστά την οδηγία. Ο κανονισμός αυτός είναι πολύ φιλόδοξος γιατί θέλησε να εισάγει μια νέα στρατηγική δραστήριου και προληπτικού χαρακτήρα, εξαιρετικά ε, ισχυρού, προωθώντας ε, το ε, προστασία από το σχεδιασμό και εξορισμού, δημιουργώντας μια νέα φιγούρα που δεν αναφέραμε αλλά που σίγουρα θα έχει μεγάλη σημασία, που είναι η υπεύθυνη προστασίας δεδομένων, αλλά και ενίσχυση της ε, στρατηγικής καταστολής, διότι θεσπίζεται ένα νέο κοινό καθεστώς κυρώσεων, ενισχύονται οι εθνικές αρχές, αλλά και οι ευρωπαϊκές αρχές εποπτείας, που έχουν αυθύνη σε αυτό το τομέα και θεσπίζονται και δεν μπορούμε αυτό να το ξεχνάμε. Σήμερα δεν, το, δεν μας απασχόλησε αρκετά μηχανισμοί εναρμόνισης αυτής της οδηγίας με νέα μέσα για συνεργασία σε θέματα έρευνας και μια νέα διαδικασία συνοχής που ακριβώς καλείται να εγγυηθεί αυτή την ευρωπαϊκή εναρμόνιση στην πράξη απέναντι στο τεχνολογικό τσουνάμι, νέα δικαιώματα και νέες εγγυήσεις ε, συγκεντρώνονται σε αυτό το κανονισμό και επηρεάζουν συγκεκριμένα παιδεία και συγκεκριμένα δικαιώματα τόσο του παιδιού όσο και νέα δικαιώματα όπως η διαφάνεια, η λύθη, το δικαίωμα στη λύθη και σίγουρα σήμερα είδαμε σαφώς πόσο υπάρχουν λανθάνουσες ανησυχίες που δεν έχει καλύψει ο κανονισμός αυτός. Μία από αυτές τις ανησυχίες είναι ακριβώς η μεταγραφή στο εθνικό επίπεδο με τους εθνικούς κανόνες, δηλαδή που, ε, νόμους που θα μετατρέψουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία σε εθνική. Επίσης έχει να κάνει με τις ασυμμετρίες που θα συνεχίσουν να υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο παρά το ότι έχουμε να κάνουμε με ένα νέο νομικό μέσο όπως ο κανονισμός Πολλές χώρες, πολλές εθνικές ε, νομοθεσίες έχουν χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες εξαίρεσης που δίνει ο κανονισμός σε πολλά θέματα και συγκεκριμένα σήμερα διαπιστώσαμε αυτό που αφορά την ηλικία συγκατάθεση των ε, ανηλίκων. Υπάρχουν επίσης ανησυχίες που αφορούν την ανάγκη συνεκτικής και ομοιογενούς ερμηνείας του κανονισμού και της ανάγκης πραγματικής και αποτελεσματικής εφαρμογής του κανονισμού. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της, ε, του enforcement, ε, του συστήματος ε, οικονομικών κυρώσεων που προβλέπεται από τον ίδιο τον κανονισμό και που επηρεάζει την επεξεργασία των δεδομένων σε διάφορους τομείς Μόλις αναφερθήκαμε στο τομέα της έρευνας, της βιοιατρικής προβληματισμοί τους οποίους θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη εμείς οι νομοθέτες γιατί θα κληθούμε να δώσουμε απαντήσεις σε αυτές τις αμφιβολίες και σε αυτές τις προκλήσεις που δημιουργούνται και θα πρέπει επίσης να δώσουμε απαντήσεις στις ανεξάρτητες αρχές προστασίας των δεδομένων. Όμως, με την εφαρμογή του κανονισμού έχουμε και λόγους να ενθουσιαζόμαστε και να ε, παροτρινθούμε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτή τη νέα νομοθεσία ε, συνεχίζει να αποτελεί την αναφορά ε, παγκοσμίω και μάλιστα στον τομέα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και μάλιστα το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής προσωπικής ζωής θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε όλα αυτά να μεταφραστούν σε πραγματικότητα, ώστε οι διεθνείς εταιρείες ε, και οι βορειοαμερικανικές κυρίως θα χρειαστεί να εφαρμόσουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα στις πολιτικές τους. Και το ίδιο και οι υπόλοιπε ήπειροι θα ακολουθήσουν με παρόμοιες νομοθεσίες. Γίνεται λοιπόν μια παγκοσμιοποίηση αυτού εδώ του νομοθετήματος. Άρα λοιπόν δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με ένα ευρωπαϊκό νομοθέτημα, το οποίο πρέπει να εφαρμόσει κάθε κράτος ένωσης. Πρόκειται για έναν κανονισμό που έχει ε, οικουμενική ε, διάσταση και γι' αυτό θα πρέπει να αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Επειδή οι συνάδελφοι αρχίζουν να φεύγουν, σας ευχαριστώ πολύ κύριο Κάγιο, ε, Ράγιο Λομπάρτε. Θα ήθελα απλά να αναφέρω και να αναφέρω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι αυτό το βήμα είναι το πρώτο βήμα στον εξυγχρονισμό του Ευρωπαϊκού Συστήματος ε, νομικού συστήματος για την προστασία των δεδομένων, αλλά έχουμε και το κανονισμό για το e-privacy που είναι υποδιαπραγμάτευση. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε καλή σχέση μαζί σας, τα εθνικά κοινοβούλια, καθώς εξετάζουμε αυτά τα πολύ σημαντικά νομοθετήματα. Η σημερινή μας διάσκεψη χαρακτηρίστηκε και από τις δικές σας συμβολές και που δείχνει πως τα κάτι μέλη δεν θα μπορέσουν να τηρήσουν τις προθεσμίες για τη μεταγραφή όλα. Ε, πρέπει να παρακολουθούμε λοιπόν την κατάσταση πολύ προσεκτικά και φυσικά καλούμε την Κομισιόν να προβεί στα απαραίτητα βήματα ώστε να μεριμνήσει για τη σωστή εφαρμογή του συνόλου της δέσμης μέτρων. Πάντως εσείς ε, βοηθήσατε στο να τονίσουμε αυτές τις ανησυχίες αλλά και τις ευκαιρίες που προσφέρει η δέσμη αυτή μέτρο. Ήταν πολύ καρποφόρα μέρα για μας το Ευρωκοινοβούλιο και την Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ και πάλι λοιπόν τους εθνικούς βουλευτές για τις εξαιρετικές σας συμβολές. Ευχαριστώ επίσης τους ομιλητές μας.